Το πρώτο τμήμα της συνεδρίασής μας είναι οι πληροφορίες που θα σας δώσω σχετικά με τη συνεδρίες των συντονιστών χθες. Εγκρίθηκε η πρόταση να γίνει γνωμοδότηση για την έκθεση της Επιτροπής Μηχανίας για την απλούστευση και την εφαρμογή των προγραμμάτων πλαισίων για την έρευνα. Η ομάδα ΕΛΚ θα κάνει την έκθεση αυτή ο κύριος Αλντι Πατριτσέλο, εισηγητής. Εγκρίθηκε μια νέα έκθεση πρωτοβουλίας για την αποτελεσματική χρήση των πιστώσεων της Ένωσης σε θέματα αποδόμησης πυρηνικών σταθμών στις νέες χώρες μέλη. Ο κύριος Μαρινέσκου, ΕΛΚ, εισηγητής. εγκρίθηκε το σχέδιο ερωτηματολογίου για τους νέους υποψήφιους του ελεγκτικού συνεδρίου Ολλανδίας Κύπρο και εγκρίθηκε και το χρονοδιάγραμμα μπορείτε να το δείτε είναι από τον Ιούνιο του 10 μέχρι τον Ιανουάριο του 2011 η Αγιάλα Σέντερ ε, εισηγείται ομάδα σοσιαλιστών επίσης εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα για την παρουσίαση της νέας ετήσιας έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου θα υποβλη... παρουσιαστεί επίσημα στην Επιτροπή την 3η 9 Νοεμβρίου. 5 Οκτωβρίου επίσκεψη στο ελεγκτικό συνέδριο όλοι οι βουλευτές της Επιτροπής καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή αν ενδιαφέρονται για να οργανώσουμε καλά την επίσκεψη αυτή. Εγκρίθηκε το τελικό πρόγραμμα της αντιπροσωπείας που θα πάει στην Κροατία και το χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη έκθεση απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αστυνομίας. Η διαδικασία θα είναι τον Ιούλιο του 2010. Αρχίσαμε επίσης να οργανώνουμε και τις αντιπροσωπείες για την Ουγγαρία ποιοι θα πάρουν μέρος, τα ονόματα, από, έριψαν την αίτηση του κ. Αντί να ζητηθεί από τις νομικές υπηρεσίες σχετικά με τον τι έλεγχο μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο στα άλλα θεσμικά όργανα. Έτοιμα οντί. Εν μέρη ενέκραναν οι συντονιστέ το αίτημα Ριβελίνη προσφυγή στι νομικέ υπηρεσίε του Κοινοβουλίου για θέματα σχετικά με τις αλλαγές που προτείνονται στο δημοσιονομικό κανονισμό. Εγκρίθηκε η πρωτοβολία να καταγραφεί στο Europarl η τελική ψήφος στην απόφαση για την απαλλαγή και όχι η ψήφος για επί του ψηφίσματος. Επίσης θα αποσταλεί επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου προτείνοντας κάθε φορά που θα έχουμε ψήφο απαλλαγή στο Κοινοβούλιο να στέλνετε επίσημη πρόσκληση σε όλα τα θεσμικά όργανα των οποίων η παρουσία κρίνεται αναγκαία. Τέλος, τροποποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής μας και θα σας αποσταλεί σε όλους σας. Αυτά για τη χθεσινή συνεδρίαση των συντονιστών. Αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχόλια... Ας περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της σημερινής συνεδρίασης που είναι η κοινή ακρόαση των Επιτροπών Προπολογισμού, Ελέγχου Προπολογισμού σε σχέση με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, όλους τους παρόντες. Αγαπητέ Πρόεδρε Χάουγ, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, τονίζω τη σημασία της σημερινής συνάντησης σε σχέση με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για κάτι που αφορά μόνο τους ε, τεχνικούς και τους υπάγγελους. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την πολιτικοθεσμική ζωή των οργάνων της Ένωσης και για όλους τους φορολογούμενους. Αυτό ισχύει κατά μείζονο λόγο σήμερα, όπου υπάρχουν χώρες της Ένωσης, που όπως ξέρετε βρίσκονται σε βαθιά δημοσιονομική και οικονομική κρίση. Πώς δαπανώνται λοιπόν τα κονδύλια της Ένωσης. Είναι ένας από τους κύριους λόγους για να έχουμε μια υγιή αποτελεσματική οικονομική ανάπτυξη. Να μειωθεί η ανεργία και να μην υπάρχουν από τη μια μεριά σπατάλες λόγω ανικανότητας των πολιτικών να διαχειριστούν τα κοινωτικά κονδύλια και από την άλλη μεριά όπως συχνά βλέπουμε από στοιχεία που μας δίνουν οι χώρες μέλη από ελέγχους της Όλαφ ή από ελέγχους του ελεγκτικού συνεδρίου υπάρχουν ακόμα και απάτες και διαφθορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού έχει σημαντικό πολιτικό ρόλο. Ελέγχει κόστος και όφελος σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μπορεί τα κονδύλια να δαπανώνται μεν, αλλά πρέπει να δούμε τι είδους προγράμματος, δημοσίου προγράμματος, χρηματοδοτήθηκε με, προγρα... με κονδύλια της Ένωσης και ήταν σκόπιμο να γίνει αυτό ή όχι. Μπορεί να είναι χρήσιμο το έργο, αλλά δεν έχει καμία κοινωνική ή πολιτική ή άλλη αναγκαιότητα σε σχέση με τα χρήματα του φορολογούμενου. Κάτι άλλο για τη σημερινή συνάντηση εξίσου σημαντικό. Μπορεί από εδώ να βγουν προτάσεις για να πετύχουμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην απλούστευση των κανόνων, μείωση της γραφειοκρατίας, που όλοι τη θέλουμε, και την ανάγκη ελέγχων. όσο πιο μικρότερη η γραφειοκρατία από μια μεριά είναι αναγκαίο. Από μια άλλη μεριά είναι αναγκαίο να έχουμε πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Λέμε πάντα ανοχή μηδέν έναντι της σπατάλης του δημοσίου χρήματος, έναντι των απατών, έναντι της διαφθοράς. Διαφάνεια, αποδοτική χρήση των κονδυλίων. Έχει εγκριθεί πρόσφατα η τεθεί σε ισχύ μάλλον η συνθήκη της Λισαβόνας που ενισχύει τις εξουσίες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας, ιδιαίτερα το δημοσιονομικό κανονισμό. Άρα έχουμε περισσότερες υποχρεώσεις και στα κράτη-μέλη. Με πικρία διαπιστώνω ότι η πρόταση της Κομισιόν την είχαμε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Αυτό βέβαια δεν διευκολύνει τις σημερινέ μας εργασίες και γενικά τις εργασίες της Επιτροπής μας. Ένα από τα κύρια θέματα για τα οποία η σημερινή μέρα θα μπορούσε να δώσει στοιχεία περισυλλογής είναι το πώς να βελτιώσουμε τον έλεγχο, το audit, έλεγχο της Κομισιόν, τον έλεγχο της Όλαφ. Χθες με την ακρόση του Επιτρόπου ΜΕΤΕ για το πρόγραμμά του τονίσαμε τη σημασία για μας της ενίσχυσης της Όλαφ και επειδή το 80% των ευρωπαϊκών κονδυλίων τα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη με τη λεγόμενη συνοδό διαχείριση, δηλαδή ουσιαστικά την κάνουν τα κράτη-μέλη και σε μερικές χώρες μέλη περιφέρειας, αλλά την τελική ευθύνη, την πολιτική την έχει η Κομισιόν. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι τι ευθύνη έχουν τα κράτη-μέλη. Χθε ρώτησα τον Επίτροπο Σεμέτα και δεν μου απάντησε. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα πάρουμε μια πιο συγκεκριμένη απάντηση εκ μέρους κάποιου άλλου από την Κομισιόν. Τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν τη στιγμή που ακόμα χώρες μέλη συνεχίζουν να παραβιάζουν σοβαρά όσον αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όσον αφορά τη διαφθορά, όσον αφορά τη δίσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στη χρήση του δημοσίου χρήματος, και είδους κυρώσεις σκοπεύει να εφαρμόσει η Κομισιόν έναντι αυτών των κρατών που ε, υποτροπιάζουν. Εμείς στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού ε, ζητήσαμε να μπει η εθνική δήλωση διαχείρισης ακριβώς σε σχέση με τις κυρώσεις στην περίπτωση που δεν τηρούνται, τηρείται η νομοθεσία. Δεν αρκούν όμως δηλώσεις αρχών γενικόλογες. Πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες. Γιατί όταν μιλάμε για δημόσιο χρήμα, δεν μιλάμε μόνο για χρήματα των οργάνων της Ένωσης, μιλάμε για τα χρήματα που προέρχονται από όλους τους φορολογούμενους. Και το κύριο των ευρωπαϊκών οργάνων θα μετρηθεί με τη διαφάνεια, με την αποτελεσματική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων των 27 κρατών μελών. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας σήμερα και δίνω το λόγο στη συνάδελφο Χάουγκ αντιπρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών για μια εισαγωγή εκ μέρους της. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω όλους ε, θερμά εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η δημόσια ακρόαση που κάνουμε σήμερα μαζί με την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών έχει σαν σκοπό να τονίσει το ρόλο μας ως συνομοθέτες στον δημοσιονομικό κανονισμό και να τον διευκολύνει αυτό το ρόλο. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις σε σχέση με το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πρόταση της Επιτροπής ή δυνατόν ούτως ώστε να υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με το δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό το οποίο μας έχει παρουσιάσει η Επιτροπή, μας έχει υποβάλει η Επιτροπή και αυτό που σήμερα ειδικά θέλουμε να συζητήσουμε σχετίζεται άμεσα με την απλούστευση του δημοσιονομικού κανονισμού. Επιθυμούμε τα χρήματά μας ε, να καταλήγουν στον πολίτη κανονικά βεβαίως αλλά και χωρίς καθυστερήσεις. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών έχει βεβαίως ε, κάθε ενδιαφέρον η διαδικασία αυτή να γίνεται σωστά. Αλλά όλοι μας από κοινού έχουμε και το συμφέρον να μην ε, υπάρχουν επιπλέον δυσχέρειες από τα άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού ε, ε, η Κομισιόν έχει αλλάξει τα μισά. Την, τελε... την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, ε, μας υποβλήθηκε το τρίτο τμήμα των προτάσεων ε, τροποποίησης και έχουμε η Κομισιόν μας παρουσιάζει τη νέα της ε, μεθοδολογία και ταυτόχρονα η Κομισιόν ε, μας ε, γνωστοποιεί και είναι το δικαίωμα πρωτοβουλίας που έχει ότι θέλει να προβεί στην αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού σε τρία τμήματα. Έχει λοιπόν κάνει υποβάλει τις προτάσεις της όσον αφορά τις αναγκαίες αλλαγές που προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και στη συνέχεια έκανε τις προτάσεις που προκύπτουν για την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και την περισμένη Παρασκευή μας παρουσίασε το τρίτο τμήμα που αφορά στην απλούστευση ακριβώς. Και αυτοί οι τρεις σκοποί θα γίνουν αντικείμενο μιας ξεχωριστής επεξεργασίας αφενός και αφετέρου εφόσον η νομοθετική διαδικασία ε, για αλλαγέ που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας εφόσον επίκειται η αλλαγή ενός άρθρου ε, αυτό επηρεάζει την ε, παράλληλη συνονομοθετική διαδικασία όσον αφορά την, ε, σε σχέση ακριβώς με την απλούστευση. Θα έλεγα, δηλαδή, ποια νομοθεσία προηγείται, για παράδειγμα, και νομίζω ότι η συγγήτριά μας έχει πάρα πολλά πράγματα να έχει, έχει να κάνει εδώ και ελπίζω ότι δεν θα χάσει την υποπτία και θα μπορεί να μας ενημερώνει τακτικά. Βεβαίως από την άλλη ε, γνωρίζουμε ότι οι αλλαγές που είναι αναγκαίες, δηλαδή όλα όσα έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας, θέλουμε να εμείνουμε σε αυτά γιατί εάν το Συμβούλιο δεν θέλει να διαπραγματευτεί μαζί μας, δεν θα υπάρξει μια αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού υπό την έννοια των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε σε σχέση με το δημοσιονομικό κανονισμό και ε, γι' αυτό θέλουμε, ε, θελήσαμε να οργανώσουμε από κοινού την ακρόαση αυτή μαζί με την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών και θα ακούσουμε τις ε, δηλώσεις του αρμόδιου επιτρόπου, του Γιάννου ε, Λεβαντόσκη. Έχουμε εδώ εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και εμπειροκνόμενους από τις διάφορες χώρες μέλη και Επίσης έχουμε ένα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου εδώ, το οποίο θα μας παρουσιάσει επίσης τη δική του άποψη. Τώρα θα ξεκινήσουμε με την εισαγωγή που θα μας κάνει ο Γιάννης Λεβαντόφσκι, ο αρμόδιος επίτροπος του προπολογισμού και στη συνέχεια θα έχουμε τις, ε, τρι, τους τρεις συγγνώμη, εμπειρογνώμονες από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και στη συνέχεια ασφαλώς θα έχουμε ένα γύρο συζήτησης στο πλαίσιο το οποίο θα τοποθετηθούν θα, κάποιες ερωτήσεις. Δεν είναι καλό. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει οι συνάδελφοι, ότι και αν πιστεύει ο Επίτροπος, να συμμετάσχουν σωστή αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού. Θα πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη δυνατή παράδοση να συζητάμε τις ε, πολύπλοκες τροποποιήσεις ε, υπομορφή μιας δημόσιας ακρόασης. Είναι καλή η παράδοση αυτή. Είμαι ευγνώμων προς τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Γνωρίζω ποια ήταν η δική σας συμβολή ε, υπό την ηγεσία της κυρίας Γκρέσλε θα σας παρουσιάσω τις βασικές κατευθύνσεις ε, της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού. Είναι η τρίτη. Η πρώτη ήταν μια τεχνική προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνας. Η δεύτερη ήταν η προσαρμογή που έχει να κάνει με την ε, ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης που συνδέεται και με την αναθεώρηση του καταστατικού των υπαλλήλων και τώρα έχουμε την λεγόμενη ετήσια αναθεώρηση, η οποία θα πρέπει να γίνεται κάθε τρία χρόνια. Εμείς προτείνουμε να μην υπάρχει υποχρέωση να γίνεται η αναθεώρηση αυτή, να γίνεται εφόσον είναι απαραίτητο. Ως προς το χρονοδιάγραμμα. Ναι, τελευταία στιγμή έγιναν όλα αυτά. Η προθεσμία ήταν αυτή τη βδομάδα, αλλά το δικό μας χρονοδιάγραμμα ε, συγκρόταν με το δικό σας. Έπρεπε να γίνουν ε, διυπηρεσιακές ε, διαβουλεύσεις για να υπάρχει ένα τελικό προϊόν το οποίο να υιοθετηθεί ε, την προηγούμενη εβδομάδα από το Σώμα των Επιτρόπων για να ε, παρουσιαστεί σήμερα εδώ. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο όλο πλαίσιο. Η αναθεώρηση γίνεται με βάση δημόσια διαβούλευση του 2009. 12 ερωτήσεις στέθηκαν, πολλές ε, απαντήσεις είχαμε αυτό, αυτές ε, κυρίως έχουν ε, να κάνουν με τις απλοποιήσεις για τους μικρούς αποδέκτες. Δεδομένης της διαδικασίας της συναπόφασης ε, που είναι χρονοβόρα, έχουμε εδώ μια σειρά κανόνων για τις επόμενες δημοσιονομικές πρόπτικες από το 2012 και μετά. Πρόκειται λοιπόν για τη βάση για την για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Προτού λοιπόν να μιλήσουμε για, πόσο, για το πόσο, ε, προτού μιλήσουμε για το μέλλον των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών, ε, θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς. Και στο επίκεντρο της προσοχής μας είναι οι κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίοι όμως δεν αποτελούν το τέλος της ιστορίας μας, όπως μας δείχνει η εμπειρία μας. Πολύ συχνά τομεακοί κανόνες είναι οι πιο σημαντικοί για τους αποδέκτες, οι οποίοι όμως αποκλίνουν από το γράμμα και από το πνεύμα του δημοσιονομικού κανονισμού. Σημαντική λοιπόν είναι η συμμόρφωση των τομεακών κανόνων με τους γενικούς κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού που είναι σαν το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός λοιπόν είναι ένα από του βασικούς μας στόχους. Ας προχωρήσουμε στι βασικέ στις βασικές κατευθύνσεις της ε, αναθεώρησης Ήταν πολλή δουλειά η αναθεώρηση πάνω από 100 ε, άρθρων από τα 187 συναλλικά ε, στον δημοσιονομικό κανονισμό που ισχύει ακόμα. Τρεις βασικές κατευθύνσεις έχουμε. Απλοποίηση. Αυτό φαίνεται και από την δημόσια διαβούλευση. Δεύτερον, τη μόχλευση και την συλλογή, την συγκέντρωση των πόρων. Διότι οι περιορισμοί, οι προϋπολογιστικοί περιορισμοί θα ε, συνεχίσουν να υπάρχουν στο μέλλον όπως και τώρα. Θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε το αποτέλεσμα της μόχλευσης και όσον αφορά τους κοινοτικούς πόρους και τους εθνικούς και τους ιδιωτικούς. Επίσης θέλουμε αυξημένη υποχρέωση λογοδοσίας όπως αφέρθηκε από τους Προέδρους των Επιτροπών Προϋπολογισμού και Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Το 80% του προϋπολογισμού εκτελείται στα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική υποχρέωση λογοδοσίας και αυτό ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες του ελεγκτικού συνεδρίου ε, με την προσδοκία να ε, πετύχουμε την πρώτη θετική ε, δήλωση διασφάλισης. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα είναι η πρώτη θετική τέτοια δήλωση. Απλοποίηση πρώτα. Θα έλεγα ότι πρόκειται για επανάσταση ε, διανοητική. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι έλεγχος των τιμολογίων. Εξετάζουμε δηλαδή περισσότερα τα εισερχόμενα παρά τα εξερχόμενα. Τι είναι λοιπόν απαραίτητο εδώ. Είναι απαραίτητο να αλλάξουμε τον τρόπο δουλειάς μας για να συγκεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα. Η απλοποίηση όμως δεν μπορεί απλά να είναι ένα σύνθημα για να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας όσον αφορά τον λογιστικό έλεγχο και τον τρόπο που εργαζόμαστε με το δημοσιονομικό κανονισμό. Έχουμε τα, εφάπαξ ποσά, ε, ε, ε, τα, τα εφάπαξ ποσά, τα σταθερά ποσοστά. Θέλουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να καταργήσουμε το πλαφόν για τα εφάπαξ ποσά. Θέλουμε επιβεβαιωμένα ιστορικά στοιχεία ε, για τους ε, αποδέκτες και να ε, εξετάζουμε τα στοιχεία αυτά και να δίνουμε αντίγραφα των σχετικών εγγράφων στις Επιτροπές Προϋπολογισμού και Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Πολλοί αποδέκτες είναι υπέρ του κλασικού καθεστώτος δαπανών, αλλά όσον αφορά τους μισθούς ε, υπάρχει το μέσο κόστος. Θέλουμε λοιπόν να εισάγουμε ένα νέο καθεστώς αντί για το καθεστώς των εφάπαξ ποσών στον νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Βλέπουμε και πάλι εδώ τα αποτελέσματα της ε, δημόσιας διαβούλευσης. Δεν είναι πια απαραίτητο να υπάρχει ε, λογαριασμός τραπέζης για τις προκαταβολές. Αυτό έχει να κάνει και με ε, τα, τους τόκους και τα κέρδη, την ανάκτησή τους Υπάρχει, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, υπάρχει όμως περιθώριο βελτίωσης εδώ πέρα ε, ως ανταπόκριση στι στις απαντήσεις της δημόσιας διαβούλευσης. Ε, από 25.000 σε 50.000 ευρώ ε, αλλάζει το κατόφλι για τις ε, χαμηλές επιχορηγήσεις. Αλλάζει και η διαδικασία και θα τροποποιήσουμε και τα κατόφλια για τις δημόσιες προμήθειες. Όσον αφορά τις, ε, την επιβράβευση και εδώ θα αλλάξουμε τους κανόνες, όλα αυτά ε, είναι κινήσεις για απλοποίηση ε, ως απάντηση στη δημόσια διαβούλευση. Δεδομένων όμως των περιορισμών στην Ευρώπη μετά την κρίση και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας. Ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό και να βελτιώσουμε ε, τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα Trust Funds της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει μέχρι 50% της χρηματοδότησης των ε, κάποιων φορέων όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα ε, και το, τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν είναι ορατή η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιος άλλος διαχειρίζεται τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει να μπορούμε να δημιουργήσουμε δικά μας trust fund αυτό είναι επίγον θέμα ιδιαίτερα στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Μας ενδιαφέρει ε, να είναι ορατές οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό που απαιτείται σήμερα όμως είναι καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί μέλος της οικονομικής οικογένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γι' αυτό εξετάζουμε τις διαδικασίες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να πετύχουμε μόχλευση. Ε, εξετάζουμε, τις, ε, εξετάζουμε νέες μορφές ε, συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και κάτι που θα μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση για τους εταίρους είναι να λειτουργούν με βάση το εθνικό δίκαιο το οποίο είναι περισσότερο γνωστό στους ιδιωτικούς εταίρους στα κράτη-μέλη. Τα θεσμικά όργανα, αλλά τα ενδιαφέρει, λιγότερο όμως ενδιαφέρει τον εξωτερικό κόσμο, ε, τα ενδιαφέρει λοιπόν να μπορούν να λάβουν δάνεια για την ε, απόκτηση κτηρίων. Ε, χρηματοδοτούμε κτίρια, αγορές κτηρίων ε, είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με την αποταμίευση όσον αφορά την κίνηση προς ε, καλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας. Είναι δύσκολη η ιστορία αυτή δεδομένων των διαφορετικών καθεστώτων στα κράτη-μέλη όπως όμως ε, πολύ σωστά τονίστηκε από τους προέδρους ε, των Επιτροπών Προϋπολογισμού και Ελέγχου του Προϋπολογισμού δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιο περιθώριο λάθους. Ε, το οποίο ε, συχνά μπορούμε να το ονομάζουμε μέχρι και διαφορά. Στην εκτέλεση, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι είμαι υπεύθυνο εγώ, ξέρω ότι το σώμα των επιτρόπων είναι οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του προπολογισμού. Θέλουμε όμως να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, πώς λοιπόν να βελτιώσουμε την ε, υποχρέωση λογοδοσίας. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο επίπεδο πολιτικών δηλώσεων. Δεν είναι εύκολος τρόπος αυτός να πείσουμε ε, κράτη-μέλη με ομοσπονδιακή δομή δεν θα ακολουθήσουν τον δρόμο των πολιτικών δηλώσεων. Γι' αυτό Θέλουμε να μεταφέρουμε στις, στον τομέα της συνοχής ε, τις δομές των γεωργικών πληρωμών. Οι, οι λοιπόν που πληρώνουν στον τομέα της συνοχής ε, θα εκδίδουν δηλώσεις διαχείρισης ε, που θα υποβάλλονται σε εξωτερικό λογιστικό έλεγχο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκπονούν συνθετικές εκθέσεις ε, για τις ε, δηλώσεις διαχείρισης. Ε, αυτό δεν είναι το τελικό βήμα και ξέρω ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Πρέπει να λάβω υπόψη όμως τις διάφορες, τα διάφορα καθεστώτα και τις διάφορες απαντήσεις που έχουμε λάβει από τα κράτη-μέλη. Αυτή λοιπόν είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Είναι σημαντικό αυτό για τις υπηρεσίες που κάνουν τις πληρωμές ε, όσον αφορά τον κίνδυνο και τις ε, κατηγορίες για διαφθορά. Ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο όμως ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο και το, ε, λογιστικό, το ελεκτικό συνέδριο ε, είναι η ε, εξέταση των προκαταβολών της ε, χρηματοδότησης ε, εκ των προτέρων. Θα πρέπει τακτικά να γίνεται εκαθάριση των ποσών αυτών. Είναι κατανόητο αυτό. Ποιο είναι το ανεκτό περιθώριο λάθους. Το θέμα εδώ δεν είναι η ανοχή του λάθους, αλλά Ε, στο κράτος μέλος που γνωρίζω εγώ καλύτερα ε, είχαμε δυσκολίες να πείσουμε τον κόσμο ότι για κάποιους τομείς ενδείκνυται υπάρχουν ε, αναλύσεις κόστους όφελους που όμως ε, παρουσιάζουν διαφορετικό περιθώριο λάθους, 2-3% ε, μπορεί αυτό να διαφέρει από τομέα σε τομέα. Ακόμα και το κόστος του λογιστικού ελέγχου είναι μερικές φορές τόσο ψηλό σε σχέση με το όφελος του λογιστικού ελέγχου που θα πρέπει να εισάγουμε την έννοια της ανάλυσης κόστους όφελους ε, στους λογιστικούς ελέγχους ε, και στην εφαρμογή γενικά. Βέβαια, όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο του διαλόγου μας με άλλα θεσμικά όργανα. Μετά, το επόμενο βήμα ποιο θα είναι. Ε, η κανονική νομοθετική διαδικασία, δεν έχουμε πια απόφαση. η με τις ε, προσαρμογές στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Έχουμε το Κοινοβούλιο, έχουμε την ε, Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και πρέπει να αναθεωρήσουμε τους κανόνες για την συναπόφαση με το Κοινοβούλιο. Οι κανόνες θα μπορέσουν να εφαρμοστούν μόνο μετά την υιοθέτηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Ρεαλιστική υπόθεση είναι λοιπόν ότι με βάση τις εμπειρίες μας από το παρελθόν θα είμαστε έτοιμοι το 2012 για εφαρμογή των νέων κανόνων. Και μιλάμε για τους βασικούς κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Στο... Κατά το τέλος ε, των ε, παρουσιών δημοσιονομικών προοπτικών, ε, πιο πολύ όμως αναφερόμαστε στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κανόνες προτού υποβάλλουμε το σχέδιο πρότασής μας, ε, το σχέδιο του προπολογισμού για το 2013. Αυτή ήταν ε, η εισαγωγή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ελπίζω ότι ε, ήταν αρκετά συγκεκριμένα τα όσα είπατε όπως ήθελε και ο κύριος Μαγκίστριτ ο οποίος ζήτησε πραγματικά συγκεκριμένες δηλώσεις εκ μέρους σας. Τώρα θα ακούσουμε τους τρεις πυρογνώμονες από τους μη κυβερνητικούς ε, οργανισμούς. Καταρχήν ο κύριος ε, Μακ Μίτσελ από το Volunteers του Λονδίνου και στη συνέχεια την κυρία Ιζαμπέλα Τότ από την Court Aid και μετά τον καθηγητή κύριο Μάρκου Ματίλα από την Ακαδημία της Φινλανδίας. Κύριε Μίτσελ, παρακαλώ. Και στη συνέχεια θα έχουμε μια συζήτηση. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Λέγομαι Μάρκ Μίτσελ, βλέπω για μια μη κυβερνική οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 1997 ασχολούμαι με ευρωπαϊκά θέματα χρηματοδότησης και για το Κοινωνικό Ταμείο στην Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα υπερεθνικά προγράμματα χρηματοδότησης και αυτή τη γνώση θα σας φέρω εδώ σήμερα για το πώς εφαρμόζονται συγκεκριμένα προγράμματα. Η πληροφόρηση είναι από τρεις πηγές. Από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο που ασχολείται με τα διορθωτικά ταμεία ήδη από το 1996, CSV που είναι με ένα φιλοθροπικό ίδρυμα που εργάζεται με κοινωνικά προγράμματα με θελοντές νέους, για νέους ε, αποκλεισμένους από την κοινωνία και άνεργους ένα άλλο δίκτυο και από τη δική μου οργάνωση, Corin Council, για εθελοντικές υπηρεσίες που δίνει μια περιφερειακή δράση στην Ανατολική Αγγλία. Η έκθεσή μου εστιάζεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, διαφορετικά ταμεία, αποκεντρωμένη δράση από εθνικούς φορείς και κεντρική δράση ε, από τις Βρυξέλλες. Στο Ηνωμένο Βασιλείο το Πεσέτρο μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν πρόσβαση σε διευθυντικά ταμεία, βοηθούνται από εσωτερικές αλλαγές που έγιναν στον τρόπο χρηματοδότηση του Ε.Β. Βέβαια, η μείωση των εσωτερικών κονδυλίων ε, ανάγκασε ε, τη στροφή προς άλλους φορείς. Από την άλλη μεριά είχαμε και το χρηματιστήριο το οποίο δεν πήγε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση γίνεται πιο ελκυστική παρά την ευρωσκεπτικιστική θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί πολλές φορές οι προπολογισμοί που τίθονται ξεπερνάνε κατά πολύ τις βραχυπρόθεσμους κραδασμούς. Παρά την ενδιαφέρουσα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη πηγή πληροφόρηση στο Μένο Βασίλειο ή το πώ θα γίνει πρόσβαση στι διάφορε μορφέ χρηματοδότηση όσον αφορά τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Τα αποκεντρωμένα προγράμματα τα λειτουργούν πολλά διαφορετικά τμήματα ή φορεί και η πληροφορία δεν υπάρχει μόνο σε ένα μέρο. Και φυσικά καμία υπηρεσία δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση με την Κομισιόν. Το τοπίο στο Ενωμένο Βασίλειο ποικίλει. Η Σκοτία, η Ιουαλία, η Βόρεια Ιρλανδία έχουν δικά της προγράμματα χρηματοδότηση με διαφορετικούς στόχου από ότι η Αγγλία. Στη Σκοτία, Βόρεια Ιρλανδία και η Ιουαλία μη κυβερνητικέ οργανώσει. ε, εφαρμόζουν πολύ συγκεκριμένα προγράμματα. Έπειτα τα προγράμματα εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο και στις τρεις περιφέρειες που ανάφερα υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις, προοπτική ε, και τρόπος εργασίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων και όπως τελικά και η απόδοση του προγράμματος είναι διαφορετική. Στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν εθνικά προγράμματα με στοιχεία που δεν υπάρχουν στην Αγγλία. Ο προπολογισμό η εθνική συμμετοχή είναι 2,5 εκατομμύρια στην Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Αγγλία, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια και τα υπάρχουν το σύστημα των αμέσων προσφορών. σε όλες τις περιφέρειες έχουμε ένα μείγμα συγχρηματοδότησης και προσφορών. Μερικά συμβόλαια πληρώνται ανάλογα με την απασχόληση. Υπάρχει, χρειάζεται να γίνει μια αρχική κατάθεση ποσού. Το μέγεθος των συμβολέων τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα και μη ιδιαίτερα προσβατά σε οργανώσεις το μη κυβερνητών οργανώσεων οι οποίες έτσι και δεν έχουν πάρα πολλά χρήματα. Χρειάζεται λοιπόν μια αρχική επένδυση η οποία πολλές φορές είναι δύσκολη να βρεθεί. Η πρόεδρος διακόπτει γιατί ο μιλητής μιλάει πραγματικά πάρα πάρα πολύ γρήγορα, διαβάζει πάρα πολύ γρήγορα. Οι οργανώσεις από είναι υποχρεωμένες να αποκλείσουν ευάλωτες ομάδες μία μελέτη για το νέο πρόγραμμα το SF του 2008 επιβεβαιώνει ότι η διαφοροποίηση στις προσκλήσεις προσφορές δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτών των οργανώσεων. Από στοιχεία που δόθηκαν από την Διοικητική Αρχή και το TSN, εσωτερική έρευνα, οι κύριοι φορείς είναι αυτοί που παίρνουν τα πιο πολλά συμβόλαια και το ποσοστό της χρηματοδότησης είναι λίγοι, πολύ μεγα, λίγες πολύ μεγάλες οργανώσεις. Και το, ο στόχος αυτών είναι το κέρδος. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το φαινόμενο αυτοί να παίρνουν τα πιο ευνοϊκά συμβόλαια για να έχουν απόδοση στην ε, επένδυσή τους μοιραία να αποκλείσει ορισμένου άλλου από την αγορά εργασία. Και μια ανάλυση που έκανε το TSN μεταξύ Ιουνίου του 2008 και Ιουλίου του 2009 μας δείχνει ότι το 25% της χρηματοδότησης του Κοινωνικού Ταμείου πάει στο στον δημόσιο τομέα ενώ η ιδιωτική χρηματοδότηση είναι 41%. Από τη μεριά της χρηματοδότησης του δημοσίου προγραμμάτων 39% και 35% αντίστοιχα. Δώδεκα οργανώσεις καλύπτουν περίπου το 40% όλων των συμβολέων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ωστόσο, αν και σας είπα ότι η τάση είναι να μειώνεται τα συμβόλαια, να αυξάνεται το μέγεθός τους, στην Ουαλία και στη Σκοτία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται χρόνος εθελοντών παράλληλα με τη χρηματοδότηση. Αυτό δεν γίνεται στην Αγγλία. Στην Ουαλία η Βουλή έδωσε τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης στην περίπτωση που υπάρχουν, υπάρχει δυσκολία στον τριτογενή αυτό τομέα. Ο τομέας αυτός πραγματικά έχει αυτή τη δυσκολία στην Αγγλία έλλειψη τεχνικής βοηθείας. Εξάλλου το άκαμπτο σύστημα συγχρηματοδότησης στην Αγγλία απέκλεισε την ευέλικτη χρήση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Στην Αγγλία ειδικά υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων και αποκλείονται μικρές κοινότητες ή διάφορες μικρές ομάδες να κάνουν αιτήσει. Στην Αγγλία υπάρχουν νέα περιφέρειες με προτεραιότητα όσον αφορά το Περιφερειακό Ταμείο. Η Ανατολική Αγγλία έχει προτεραιότητες μια οικονομία χαμηλού άνθρακα προκειμένου να προωθηθεί η οικονομία της γνώσης, το επιχειρηματικό πνεύμα βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά τη δέσμευση των μη κυβερνητικών οργανώσεων υπάρχουν μερικές θετικές εξελίξεις το Disability Essex παραδείγματος χάρη ε, έχει ένα, μια, ένα πρόγραμμα για βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες ενώ το South End IMCA ε, χρηματοδοτεί υπηρεσίες για νέους πολίτες στην πόλη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια κληρονομιά κατά κάποιο τρόπο υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου στην περιφέρεια αυτή. Η οικονομική διαχείριση ε, πάντως ε, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Το Περιφερειακό Ταμείο χρησιμοποιείται σε ένα όχημα ενθάρρυνσης επένδυσης κεφαλαίου. Οι περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις θέλουν χρηματοδότηση για να μπορέσουν να υποστηρίξουν την υπηρεσίες και κατάρτιση των πελατών τους. Όταν όμως χρειάζεται υποστήριξη εκ μέρους του δημόσιου τομέα και δεν υπάρχει εγγύηση για περίοδο πέραν του τρέχοντος οικονομικού έτους υπάρχει δυσκολία στη χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Ταμείο, αποκεντρωμένα ταμεία και πρόσβαση σε αυτά. Δεν έχει αλλάξει και πολύ εικόνα τον τελευταίο καιρό. Παρά το γεγονός ότι τα διαχειριστικά όργανα μπορεί να αλλάζουν, τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας του οργανισμού αυτού παραμένουν τα ίδια και ο δείκτης επιτυχίας είναι σχετικά υψηλός. Ο Εθνικός Φορέας ερμηνεύει τους κανόνες της Ένωσης στο τοπικό επίπεδο και πλαίσιο. Τα έντυπα είναι συνταγμένα με βάση το εθνικό περιεχόμενο. Η χρήση εθνικών εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση των αιτήσεων είναι επίσης ένα δεδομένο και είναι πιο εύκολο να, γίνουν, να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ των εθνικών φορέων προκειμένου να αναπτυχθούν τα αντίστοιχα προγράμματα. Κατά μέσο όρο, το 60% των αιτήσεων, όπως τα προγράμματα Grundvik, Leonardo και Youth in Action, είναι επιτυχή. Πρόσβαση σε κονδύλια άμεσα στην Κομισιόν. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον και το πιο δύσκολο σε πρόσβαση ιδιαίτερα για φορείς που δεν έχουν έδρα στις Βρυξέλλες. Πολλές φορές η γλώσσα των προσφορών δεν είναι σαφής. Η διαδικασία των αιτήσεων μπορεί να είναι περίπλοκη για τις μη κυβερνικέ οργανώσεις. Μερικέ φορές είναι δύσκολο να κάνουν την αίτηση μέσω ίντερνετ. Θέμα γλώσσας, χρειάζεται πολλής χρόνος και πολλές φορές όλα αυτά οδηγούν σε αποτυχία παρά το ότι το αίτημα είναι καλής ποιότητας. Αν και οι γενικέ διευθύνσει δίνουν χρόνο 6 εβδομάδων, μερικές φορές ο χρόνος είναι πολύ πιο μικρός προκειμένου να ετοιμαστεί το πρόγραμμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η εθνική Συνιστός απαιτεί 12 εβδομάδες για την αίτηση. Η συγχρηματοδότηση μετρητά είναι μεγάλο θέμα για τις μη κυβερνικές οργανώσεις τα κλασικά τραστ και ιδρύματα κλπ. δεν υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έπειτα, όπω η δημόσια χρηματοδότηση περνάει σε συμβόλαια, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει δεν είναι δυνατόν να ε, ε, συμπεριλάβουν υπερσυνοριακή εργασία στο έργο τους. Η λήψη αποφάσεων καθυστερεί. Συχνά σημαίνει έξι μήνες, διάφορες καθυστερήσεις σε προγράμματα Επίσης, αν χρειαστεί να γίνει κάποια αλλαγή στην απόφαση και αυτό χρειάζεται πολύ χρόνο. Συμπερασματικά, η χρηματοδότηση εκ μέρους της Ένωσης είναι σημαντική συνιστόση για τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στα κράτη-μέλη και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Η αρχή της επικουρικότητας που σημαίνει ευθύνη για τη διαχείριση των διορθωτικών ταμείων στα κράτη-μέλη δυσκολεύει την Ένωση στο να είναι βέβαιη ότι η χρηματοδότηση θα ακολουθήσει στους στόχους της. Η Ευρώπη 2020 δεσμεύει τα κρατη στο να μειώσουν τους στόχους για τη φτώχεια και την αγορά εργασίας, αλλά δεν υπάρχει μηχανισμός που να υποστηρίζει αυτούς τους στόχους με επένδυση εκ μέρους των διορθωτικών ταμείων. Στον Ηνωμένο Βασίλειο εργαζόμαστε ιδιαίτερα με αυτούς που είναι πρόσφατα άνεργοι με μη κυβερνητικέ οργανώσει που παραδοσιακά ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Ο αποκλεισμό του χρόνου εθελοντών στη χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τα διαφορετικά ταμεία είναι απογοητευτική, διότι από ό,τι ξέρουμε αυτό το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανονισμοί, αλλά συχνά ε, είναι, απαγορεύεται λόγω εθήμων και πράξης, πρακτικής. οι απαιτήσει ελέγχου παραμένει ένα βάρο σε κάθε επίπεδο σε σχέση με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Θα πρέπει να είναι πιο αναλογική ή ανάλογα με προδιαγραφές, ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές. Όσον αφορά τα κεντρικά κονδύλια, χρειάζεται απλούστευτε τι διαδικασίε. Μια έννοια πρώτης φάση αίτηση να ελαχιστοποιηθεί η το πρώτο μέρο τη δουλειά που χρειάζεται. Αυτό θα διευκολύνει πολύ τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Πολλά από τα θέματα που ανέφερα εδώ σε σχέση με τα κεντρικά κονδύλια τα έχουν αναφέρει και άλλε μη κυβερνητικέ οργανώσει τη Βρυξέλλε. Σε σχέση με την απάντηση που δόθηκε στο δημοσιονομικό κανονισμό από την ομάδα Active Citizenship το Δεκέμβριο του 2009. Ωστόσο, ένα πρώτο κείμενο του νέου κανονισμού φαίνεται ότι ο χρόνος των εθελοντών, οι απαιτήσει ελέγχων και οι απλουστευμένες διαδικασίες ακόμα δεν έχουν ε, τύχη ε, μιας σαφούς απάντησης, σαφούς Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μίτσελ. Πράγματι μας παρουσιάσετε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών του δημοσιονομικού κανονισμού και μας ε, δείξατε ότι δεν μπορούμε να απειλήσουμε εμείς όλα από την Ευρώπη, για να το πω έτσι. Ωστόσο, μία φράση κράτησα στο μυαλό μου. Δεν όσον αφορά τη χρηματοδότηση δεν, ε, ε, δεν υπαγόμαστε σε στον εθνικό, σε εθνικά προβλήματα. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε την κυρία Τότ που είναι εμπειρογνώμων από την Court 8. Ε, δέκα λεπτά κυρία Court 8, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα προσπαθήσω να επιμικρύνω την ε, ομιλία μου. Λέγομαι Σαμπέλα Τότ, εργάζομαι για την ε, καθολική οργάνωση της Ολλανδίας για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια Court Aid και θα μιλήσω εκ μέρους της Concord που είναι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Εκπροσωπούμε 24 εθνικές ενώσεις και διεθνή ε, δίκτυα τα οποία εκπροσωπούν περίπου 1.600 μη κυβερνητικές οργανώσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κάνουμε πολλές πολιτικές ε, δράσεις και βρισκόμαστε σε ένα διάλογο με τους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς και άλλες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών το, η συνολική χρηματοδότηση στην Concord ανέρχεται σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ ανέτος και υπάρχουν περίπου 25 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ιδιώτες δωρητές που υποστηρίζουν την εργασία αυτών των μελών. Ε, χαιρετίζουμε πάρα πολύ την ευκαιρία να συμβάλλουν σήμερα στο θέμα αυτό κατά πόσο η τελευταία μεταρρύθμιση είχε κάποια αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση του, διοικητικού, του γραφειοκρατικού άχθου στο επίπεδο της αναπτυξιακής εργασίας. Και όλα αυτά βασίζονται στις ε, διαβουλεύσεις που κάναμε το 2009 με εκείνα τα μέλη που είναι ενεργά στο ε, τομέα της αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις εκτιμούν την ανάγκη ενός περιεκτικού δημοσιονομικού κανονισμού ο οποίος εξασφαλίζει τις βέλτιστες πρακτικές. Θέλουμε να έχουμε προγράμματα υψηλής ε, ποιότητας που σέβονται το δημοσιονομικό κανονισμό και είναι υπόλογα στους προς τους Ευρωπαίους φορολογούμενους καθώς και στις ε, ε, στους δήμους και τις κοινότητες που εξυπηρετούμε και που δέχονται αυτά τα χρήματα. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε πολλά διοικητικά βάρη. Έχουμε συνείδηση ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά ε, θέλουμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας και ε, λογοδοσίας. Επίσης, μια αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού δεν θα πρέπει να αυξήσει το διοικητικό φορτίο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ούτε να επιφέρει πλέον εμπόδια τα οποία θα μειώσουν την αποτελεσματικότητά μας. Υπερβολικός έλεγχος μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα και να αποθαρρύνει τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των κοινωτικών κονδυλίων. Κάθε αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί βάσει των αρχών της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Επίσης θεωρούμε ότι όλες αυτές οι αρχές είναι εξίσου σημαντικές μετά από την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας αναγνωρίζουμε ότι η παρούσα αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστεί στο νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή του προϋπολογισμού που ευθυγραμμίζεται με τη νέα συνθήκη και την εντολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Υπό την έννοια αυτή η Concord συμφωνεί και υποστηρίζει το ε, το, συνέδριο των, ε, το ελεγκτικό συνέδριο, τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά τη σημασία της ε, ενίσχυσης της ευθύνης, της λογοδοσίας και της ποιότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης στο επίπεδο των αντιπροσωπιών θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει οι οργανωτικές δομές των αντιπροσωπιών της Ένωσης να τεθούν ε, σε κίνδυνο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με, την, με τις άμεσες επιχορηγήσεις των τοπικών οργανώσεων στον τομέα αυτό, στις αναπτυσσόμενες χώρες ειδικότερα. Τώρα θα κάνω ορισμένε παρατηρήσει όσον αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό και του κανόνε εφαρμογή. Καταρχήν, ε, ε, θα τα διατρέξω εντάχει, αν μου επιτρέπετε, θα πω κάποια πράγματα για τις επιχορηγήσεις. Η γενική εκτίμηση είναι το παρόν σύστημα για την ε, κοινοποίηση της ε, πρόσκλησης υποβολής προσφορών, λειτουργεί καλά. Ωστόσο, προϋποθέτει μια καλή κατανόηση του συστήματος ε, που ορισμένε οργανώσει δεν διαθέτουν, ιδιαίτερα οι εταίρε μα στι αναπτυσσόμενε χώρε. Η Concord χαιρετίζει τι βελτιώσει που έγιναν του τελευταίου μήνε του 2009 με την ε, δημοσίευση των ετήσιων προγραμμάτων online για θεματικά και γραφικά προγράμματα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην μελέτη που έκανε η Concord, σε σχέση ακριβώς με τις προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, υπάρχουν κάποιες ε, αποκλίσεις όσο, όταν δημοσιεύονται οι προσκλήσεις υποβολή προσφορών στο επίπεδο των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα την ε, συγχρηματοδότηση, τα μέλη της Concord υποστηρίζουν την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας της απαιτήσεις για τη συγχρηματοδότηση. Ε, περισσότερη ευελιξία είναι αναγκαία αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υποστηρίξει όλους τους τύπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, σε αναπτυσσόμενες χώρες και ευρωπαϊκών ε, οργανώσεων, ιδιαίτερα εκείνων των νέων χωρών μελών, που ενδεχομένω έχουν λιγότερε δυνατότητε όσον αφορά την εξέβρεση χρηματοδότηση. Οι ισχύοντε κανόνε που επιτρέπουν την συγχρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνουν. Όσον αφορά τώρα τις επιχορηγείς βάση της ε, αποδοτικότητας σε σχέση με τα καταποκοπή ποσά, τα μέλη της Concord δεν υποστηρίζουν την εισαγωγή της επιβολής ενός καταποκοπή ποσού στα, στο άμεσο κόστος μιας α, ε, δράσης. Ε, συστήνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει το ισχύον σύστημα του, της παρακολούθησης ε, γιατί θεωρούμε ότι τα καταποκοπή ποσά συνδέονται με κάποια προβλήματα και δεν επιτρέπουν την πλήρη ανάκτηση των ε, κονδυλίων. Οι περισσότερες μη κυβερνητικέ οργανώσεις αυτή τη στιγμή έχουν ε, πολιτικές που εξασφαλίζουν ότι όλες οι δαπάνες καλύπτονται, ε, ανακτώνται πλήρως και οι δωρητές συμβάλλουν με ένα σωστό, με ένα δίκαιο μερίδιο κάλυψη αυτού του κόστους. Θεωρούμε ότι η εισαγωγή του καταποκοπή ποσού θα διαστρεβλώσει αυτή την ε, πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά τις ε, πληρωμές για τις ε, εκροές, η κάλυψη του κόστου στη βάση του, των εκροών δεν είναι μια ρεαλιστική δυνατή δυνατότητα για τις επιχογυρηγήσεις γιατί ε, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Οι συστάσεις είναι το βασικό θέμα ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια απλούστευση στη διαχείριση του προπολογισμού, εξασφαλίζοντα ότι οι δαπάνε των μη κυβερνητικών οργανώσεων καλύπτονται και ότι ο δωρητή από την άλλη πλευρά, ο χορηγό, δεν πληρώνει για δαπάνε που δεν υπάρχουν πιστεύουμε ότι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στο πραγματικό κόστος αλλά μειώνει το διοικητικό άχθος με την ε, παρακολούθηση αυτών των δαπανών είναι η πιο προοδευτική ε, πολιτική. Ε, τώρα, θέλουμε επίσης να διατηρήσουμε την υπάρχουσα ευελιξία ε, όσον αφορά τα κατόφλια για, τα μικρά, για τις μικρές επιχορηγήσεις, η Concord πιστεύει ότι τα κατόφλια ε, για χαμηλές επιχορηγήσεις ορίζονται πολύ σωστά. Και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να παραμείνει αρχή του ε, θεμητού ανταγωνισμού και της μεταχείρισης μεταξύ των αποδεκτών ή των δικαιούχων των επιχορηγήσεων η διαβάθμιση των επιχορηγήσεων προς τα κάτω όσον αφορά ε, τρίτα μέρη είναι αναγκαία ορίζοντας ένα μέγιστο ποσοστό σύμφωνα με το συνολικό, συνάρτηση με το συνολικό όγκο ενός προγράμματος. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτές οι οργανώσεις δεν θεωρούνται επίσημοι εταίροι των ετούντων. Τώρα, όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσιονομικών ε, φακέλων, όσον αφορά τις ε, πληρωμές των ε, προκαταβολών, η Concord θεωρεί ότι τα επιτόκια για τις προκαταβολές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κάποιες δραστηριότητε των project ή για επιπλέον πρωτοβουλίες ή ιδέες που σχετίζονται με τη δράση αυτή. Ε, θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι οι δικαιούχοι επίσης ε, έχουν ένα μερίδιο στις προκαταβολές εφόσον οι προκαταβολές ε, περιορίζονται στο 90% της συνολικής επιχορήγησης στην περίπτωση της Europe Aid. Όσον αφορά τώρα τις εγγύησει για τις προκαταβολές, η Concord θέλει να προτείνει δύο πράγματα. Πρώτον, οι αποκλήσεις, θα πρέπει, οι εξαιρέσεις θα πρέπει να χορηγούνται στη βάση της εκτίμησης κινδύνου όσον αφορά την ελόγω οργάνωση και δεύτερον να δημιουργηθεί ένα συλλογικό ταμείο όπως έγινε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας. Ε, θα αναφερθώ εν συντομία στη γραφειοκρατία για τους ετούντες. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό σχετίζεται με τον τρόπο που οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων της Europe Aid εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή και λιγότερο στον ίδιο αφορά το λιγότερο τον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό. Ε, Πιστεύουμε ότι η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων εν γέννη έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της μεθόδου καταχώρησης Παντορ και της ε, πρώτης φάσης μιας βασικής κοινοποίησης ενός προγράμματος. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να χρησιμοποιείται μια διαδικασία σε δύο στάδια. Καταρχήν να γίνεται μια βασική κοινοποίηση και μετά να υποβάλλεται η πλήρης πρόταση. Θεωρούμε ότι όλα αυτά συνιστούν βελτιώσεις και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συστηματικά. Η Concord ε, επαναλαμβάνει το αίτημά της να χρησιμοποιούνται οι περιορισμένες διαδικασίες σαν ένας γενικός κανόνας. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η βραχία περίοδος προετοιμασίας των προτάσεων. Όσον αφορά το Παντόρ, πιστεύουμε ότι είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ήταν δύσκολο να χρησιμοποιηθεί σαν ηλεκτρονικό εργαλείο ιδιαίτερα με, για τους εταίρους μας, τους τοπικούς εταίρους, θα ιδιαίτερα δύσκολο να το χρησιμοποιήσουν ως ηλεκτρονικό εργαλείο. Ε, επίσης χαιρετίζουμε την προσπάθεια της ε, Επιτροπής προς μια τυποποιημένη μέθοδο υποβολής ε, των προσφορών. Άλλες συστάσεις της ε, Concord είναι οι εξής. Θα θέλαμε να προτείνουμε προς τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να εξετάσουν το θέμα του ΦΠΑ και της μη επιλεξιμότητας των ε, φόρων. Αυτό είναι ένα θέμα που επανέρχεται. Η Concord προτείνει η DCI και το EIDHR ε, να οι, ρυθμίσεις, οι σχετικές ρυθμίσεις να συμμορφώνονται με το να συμμορφωθούν με το παρόν κείμενο, με το φυστάμενο κείμενο του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Γιατί υπάρχει το άρθρο 172α που δεν επιτρέπει την επιλεξιμότητα των φόρων. Εμείς θα θέλαμε να υπάρξει η δυνατότητα οι φόροι και το ΦΠΑ να θεωρηθούν ε, ως ε, επιλέξιμες ε, δαπάνες γιατί και αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην διαδικασία λήψης απόφασης και αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο οικονομικό κίνδυνο. Χρειάζεται μια ταχεία επίλυση αυτού του προβληματικού θέματο, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι συμβάσει επιχορηγήσεων που έχουν υπογραφεί το 2007, περιλαμβάνοντα επίση την δυνατότητα εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων αναδρομικά. Όσον αφορά τώρα το, τις, άμεσες, τις έμεσες ε, δαπάνες, όσον αφορά τις ισοτιμίες, ο δημοσιονομικός κανονισμός δεν αναφέρει τίποτα εν σχέση με την αντιμετώπιση των ισοτιμιών. Στην περίπτωση του ε, ε, Europe Aid, ε, οι, οι δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις ισοτιμίες του Infor Euro για τη μετατροπή σε ευρώ όλων των δαπανών και αυτό δημιουργεί προβλήματα ε, σχέση, και επίσης προβλήματα ρευστότητας, κάτι το οποίο δημιουργεί επίσης και αποκλήσεις μεταξύ των πραγματικών δαπανών και των δαπανών που αναφέρονται ως δαπάνες, που δηλώνονται ως δαπάνες. Ε, θα πρέπει λοιπόν, ε, θεωρούμε, να συμπεριφθεί στο δημοσιονομικό κανονισμό και στους κανόνες εφαρμογής μία πρόταση σε σχέση με, την, με το ζήτημα του χειρισμού των ισοτιμιών. Εμείς ε, προτείνουμε τη χρήση των ε, ισοτιμιών όσοι έχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, επίσης προτείνουμε τη δημιουργία ενός ε, μηχανισμού διαιτησίας στην περίπτωση απόκλησης από τους κανόνες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διστάμενες ερμηνείες, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε οι κανόνες να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλες τις υπηρεσίες στις Βρυξέλλες και στις αντιπροσωπείες τους. Τώρα, θα έρθω στα συμπεράσματα. Επαναρχόμενοι στο θέμα κατά πόσο η τελευταία μεταρρύθμιση είχε επιπτώσει στη μείωση του διοικητικού άφου στι μη κυβερνητικέ οργανώσει που εργάζονται στον αναπτυξικό τομέα, είναι σαφέ ότι ακόμα και αν ε, δούμε ε, την πρώτη του δημοσιονομικού κανονισμού τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα τα οποία προσθέτουν ένα μεγάλο διοικητικό και τεχνικό άχθο στην καθημερινή εργασία των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να ε, προσεγγίσει αυτά τα προβλήματα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού και των κανόνων εφαρμογής. Ε, ξέρουμε ότι έχει ανοίξει η πόρτα για μια άμεση ε, συνεργασία από την Επιτροπή, αλλά παρόλα αυτά είναι τόση πολύ μεγάλη γραφειοκρατία των κανόνων που δυσχεραίνεται αυτό το έργο. Ε, ζητούμε από όλου του ενδιαφερόμενου, του εμπλεκόμενου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο να εξετάσουν τις δικές τους εισφορές όσον αφορά την επικείμενη αναθεώρηση δημοσιονομικού κανονισμού. Ε, οι συγκεκριμένε στάσει μα έχουν ω εξή: να αναθεωρηθεί ο δημοσιονομικό κανονισμό και οι κανόνε εφαρμογή, ώστε να διασφαλίσουμε μία, έναν ε, σωστό έλεγχο των ε, δικαιούχων των επιχορηγήσεων, να εξασφαλίσουμε δεύτερον την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ, τρίτον να επιτρέψουμε τη χρήση των ισοτιμιών όσα έχουν αυτή τη στιγμή, να επιτρέψουμε να αναπτύξουμε ένα γενική διεύθυνση, ένα κοινό εγχειρίδιο για όλους τους χρήστες, τόσο για τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για τους ε, δικαιούχους των επιχορηγήσεων να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό διαιτησία στην περίπτωση που υπάρχουν ε, διαφωνίες που δεν μπορούν να επιληθούν στις Βρυξέλλες, να αυξήσουμε μια κανονική κατάρτιση ε, στο επίπεδο των αντιπροσωπιών και στο επίπεδο των δικαιούχων και να έχουμε επίγνωση της ανάγκης ενός σταθερού νομικού πλαισίου για την εφαρμογή του προπολογισμού στο επίπεδο των αντιπροσωπιών της Ένωσης, ακολουθώντας ε, στη συνέχεια συγγνώμη, της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη ανάπτυξης μιας ε, δημιουργικής σχέσης μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τότ. Δεν ήταν 10 λεπτά αυτά, παραπάνω ήταν. Ε, η έκκλησή σας ε, για ισότητα όσον αφορά τις πληρωμές ε, καθώς και την ευελιξία. Νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Περνάμε πολύ γρήγορα στον καθηγητή Μάτιλα Ίσως καταφέρει αυτό πραγματικά να τηρήσει με φιλανδικό τρόπο το δεκάλεπτο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Επιτροπές Προϋπολογισμού και Ελέγχου του Προϋπολογισμού για την ευκαιρία αυτή να μιλήσω στη σημαντική αυτή ε, ακρόαση. Ε, πρόσφατα ε, η Βασιλική Εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε έκθεση ε, ο επιστημονικός αιώνας, η διασφάλιση της μελλοντική ευημερία. Ε, στην έκθεση αυτή ε, βάζει την επιστήμη και την καινοτομία στην καρδιά της στρατηγικής για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, συστήνει, συνιστά να μπουν προτεραιότητες, να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις στους, ε, στην αριστεία και στην καλύτερη ευθυγράμμιση επιστήμης ε, και καινοτομίας απέναντι στις ε, παγκόσμιες προκλήσεις. Γιατί η επιστήμη και η καινοτομία είναι τόσο σημαντικές στην οικονομία και στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό. Καταρχήν, η επιστήμη και η καινοτομία δημιουργούν νέα γνώση, μεταμορφώνουν τον τρόπο που ζούμε, δημιουργεί νέα κατανόηση, νέες βιομηχανίες, νέες θέσεις απασχόλησης και μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και τα προβλήματα. Η Κομισιόν ε, στην στρατηγική 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και ενταξιακή ανάπτυξη ε, παρουσιάζει τρεις ε, προτεραιότητες. Καταρχήν ε, την έξυπνη ανάπτυξη, την, μια οικονομία που να βασίζεται στην γνώση και στην καινοτομία. Μία από τις ναυαρχίδες στις πρωτοβουλίες αυτές είναι η Ένωση της Καινοτομίας που προβλέπει χρηματοδότηση για την ε, έρευνα και την καινοτομία ώστε να διασφαλιστούν οι καινοτόμες ιδέες οι οποίες ε, να μπορέσουν να ε, διασφαλίσουν καλύτερη ζωή, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες. Και στις άλλες πρωτοβουλίες η γνώση είναι σημαντικό στοιχείο. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για δημοσιονομικό κανονισμό στο πλαίσιο αυτό. Μιλάμε για την ελκυστικότητα της ε, του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και, την, ε, και της βασικής μορφής εφαρμογής του του 7ου προγράμματος πλαισίου ε, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και σχετικές δραστηριότητες. Η Κομισιόν θέλει να απλοποιήσει την εφαρμογή των προγραμμάτων πλαισίων για την έρευνα ε, έχει εκδώσει ανακοίνωση και το Συμβούλιο το συζητάει. Η Κομισιόν έχει προτείνει μια σειρά σημαντικών μέσων για την ε, απλοποίηση και μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε με τα περισσότερα από αυτά. Οι κοινότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας όλες υποστηρίζουν ότι αυτή τη στιγμή η, η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία είναι λιγότερο ελκυστική από την εθνική χρηματοδότηση ή τη χρηματοδότηση από άλλες πηγές. Διότι ε, συνεπάγεται τεράστια γραφειοκρατία. Το μήνυμα αυτό της ερευνητικής κοινότητας δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφές. Κάτι πρέπει να γίνει στο εγγύς μέλλον. Το επιστημονικό περιοδικό Nature πριν από κάποιους μήνες όσον αφορά την ιστορία και το πλαίσιο της κατάστασης αυτής έγραφε το εξής. Νέε κατευθυντήριε ε, γραμμέ δημοσιονομικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εισήχθησαν το 2004 και που απαιτούν αναλυτική λογιστική που δεν ε, επιτρέπει περιθώριο ε, για διαφθορά. Αυτό ήταν και ο στόχο άλλωστε. Ε, Ω αποτέλεσμα όμω, κάθε, δραχμή, κάθε λεπτό που δίνεται για κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα θα πρέπει να αιτιολογείται και πριν και μετά τη δαπάνη του. Αυτό μας φέρνει σε μια κατάσταση όπου η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και οι ε, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και προκλήσεις ε, ε, στο, στον πέρα της έρευνας δεν είναι πια ελκυστικές για αυτούς που θα έπρεπε να ενδιαφέρονται περισσότερο για την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ερευνητές υψηλού επίπεδου. Τι χρειάζεται λοιπόν. Ε, χρειαζόμαστε ε, διατάξεις ε, που να σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά μέσα χρηματοδότησης. Όσον αφορά τους κανόνες για τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος συντονισμού των κανόνων ανάμεσα στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Θα πρέπει να εφαρμόζονται στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές, στην δημοσιονομική διαχείριση και στη λογιστική. Οι καθυστερήσεις είναι επίσης ένα πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται οι καθυστερήσεις ε, στην ε, χρηματοδότηση αφού έχουν υποβληθεί όλα τα σχετικά έγγραφα και έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ε, ενός ερευνητικού προγράμματος. Αυτό πονάει ιδιαίτερα και τα πανεπιστήμια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία. Τα προγράμματα χρηματοδότησης ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας ε, αποτελούν σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας είναι ελκυστική, χρειάζεται όμως περαιτέρω απλοποίηση όσον αφορά τις ε, διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και λογιστικής. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι να παρουσιάζει την ιδέα του να ε, να καταργηθεί, να αλλάξουν οι κανόνες όσον αφορά την πρώτερη χρηματοδότηση. Ε, η απέτηση για διαφορετικό ε, λογαριασμό τραπέζης για κάθε πρόγραμμα είναι επαχθής και η διαδικασία συνεπάγεται πολλές ώρες εργασίας για μικρά χρηματικά ποσά. Οι αλλαγές που προτείνει ο Επίτροπος λοιπόν ε, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες. Υπάρχει η δήλωση των Trust Researchers ε, που υπεγράφει από πάνω από 12.000 ερευνητές ε, και που υποστηρίζει ότι οι παρούσες, ο παρόν δημοσιονομικός κανονισμός μεταχειρίζεται την έρευνα σαν να είναι διαδικασία παρόμοια με την προμήθεια αγαθών. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό για τους ερευνητές, ε, τις οργανώσεις τους, ε, ούτε και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε η ε, τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού να οδηγήσει σε ειδικού κανόνες για την έρευνα. Αυτή τη στιγμή πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι το διοικητικό άχθος είναι κάτι το οποίο ευνοεί τους ανταγωνιστές μας. Ελπίζω στο μέλλον αυτό να πάψει να ισχύει. Ο Δημοσιονομικός Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης ελπίζουμε ότι θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ε, έρευνας υψηλού επίπεδου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά Ματήλα. Πράγματι τηρήσατε με φιλανδικό τρόπο το δεκάλεπτο, μιλήσατε λιγότερο από δέκα λεπτά. Αυτό μας βοηθάει να τηρήσουμε το πρόγραμμά μας. Νομίζω ότι ήδη καταλάβαμε πολύ καλά ότι η έκκλησή σας ε, είναι να απλοποιηθούν γενικά οι κανόνες. Λέτε όμως επίσης ότι πρέπει να σκεφτούμε μήπως στον τομέα της ε, έρευνας, να σκεφτούμε μήπως στον τομέα της έρευνας θέλουμε ξεχωριστούς κανόνες. Νομίζω ότι αυτό προσεγγίζει πολύ τη θέση της εισηγήτριάς μας, διότι μας λέει ότι θα πρέπει ε, να έχουμε διαφορετικούς κανόνες ε, στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανονισμού. Ε, θα ήθελα τώρα να δώσω τη δυνατότητα στους συναδέλφους όχι να κάνουν δηλώσεις, να θέσουν ερωτήσεις. Διότι εδώ θέλουμε πραγματικά να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Ingrid Gressle πρώτη και μετά Έκλεισε το μικρόφωνο της Ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Επίτροπο. Ακούσαμε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η πληθώρα των κανόνων. Τι κάνει λοιπόν η Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού για να επηρεάσει τα ειδικά προγράμματα που θα έρθουν για τη νέα δημοσιονομική περίοδο. Γιατί ανησυχώ τα πράγματα θα συνεχίσουν όπως, όπως μέχρι τώρα. Δηλαδή ο καθένας θα κάνει ε, τα δικά του και θα ε, προσπαθούμε να επιβιώσουμε τις διάφορες αντιφάσεις έχουμε πολλά παραδείγματα ότι δεν είναι ο ίδιος ο δημοσιονομικός κανονισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία αντιβαίνουν προς βασικές αρχές που έχουμε επιβάλει στον ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Το να ασκήσει εδώ μια, κανείς μια επίδραση είναι σημαντικό, κύριε Επίτροπε. Πώς θα το πράξετε, κύριε Επίτροπε, ούτως γιατί να μην ε, μπορεί το κάθε ταμείο να κόψει και να ράψει τους κανόνες στα μέτρα του και να υπάρχουν όλες αυτές τις αντιφάσεις. Θα ήθελα πραγματικά μια σωστή απάντηση πάνω σε αυτό. Και μια ερώτηση προς τον κύριο Μίτσελ. Εάν σας κατάλαβα καλά κύριε Μίτσελ, σύμφωνα με τα όσα είπατε ε, και μας παρουσιάσετε την ε, ποικιλία που υπάρχει, την ποικιλομορφία στη Μεγάλη Βρετανία όσον όσον αφορά τα, ε, τις δαπάνες αυτές. Νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να υπάρξει μια απλούστευση ούτως ώστε το φάσμα της χρήσης των ε, κονδυλίων να περιοριστεί. Το ερώτημα είναι κατά πόσο θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα έχει νόημα στη δική σας περίπτωση. Ε, θα ήθελα την κυρία να ευχαριστήσω την κυρία Τότ για, τα, για τις συγκεκριμένες προτάσεις που έκανε. Όσον αφορά το ΦΠΑ, κύριε Επίτροπε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα με τις τρίτες χώρες, αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι δυνατόν να παραιτηθούμε από το ΦΠΑ. Όταν και πώς ε, εκτιμάνει κάτι τέτοιο όταν υπάρχουν επιδοτήσεις σε κάποια προϊόντα όσον αφορά την απαλλαγή από το ΦΠΑ. Είναι εφικτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για ο κύριο Μίτσελ ανάφερε την Ουαλία κάποιες φορές. Και ιδιαίτερα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την διαχείριση των διαφορετικών κονδυλίων. Είναι δύσκολο μικρές οργανώσεις να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά και στο παρελθόν εγκρίναμε προγράμματα, ίσως πάρα πολλά, μου τον στόχο 1, χιλιάδες προγράμματα στην Ουαλία, με ερωτηματικό. Έχουν επίπτωση στο να αυξήσουν το βιωτικό επίπεδο, να αυξήσουν το ΑΕΠ στην Ουαλία κλπ. Γι' αυτό η τάση στην Ουαλία είναι να εγκρίνει μόνο μεγάλα προγράμματα και να ζητάει από οργανώσεις να παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό για τις προμήθειες στην εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων και ρωτώ τον κύριο Μίτσελ θεωρεί ότι είναι καλύτερο εμείς να έχουμε πιο μεγάλα προγράμματα και να χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο είναι πιο εύκολο για τις μικρές οργανώσεις ή να συνεχίσουμε να έχουμε πολλές, πολλά μικρά προγράμματα. Επίσης ανάφερε ο κύριος Μίτσελ την, τον συνδυασμό της χρηματοδότησης. Έχουμε αυτό που λέμε Targeted Match Fund που είναι μια για μικρέ οργανώσει ένα τελευταίο καταφύγιο κατά κάποιο μερικές φορές όπου η χρηματοδότηση είναι πολύ πολύ μικρή και ένα τμήμα της απάντησης να δούμε την, το ρυθμό παρέμβαση, το ποσοστό παρέμβαση, Να το σχολιάσει αυτό ο κ. Μίση. Ένα άλλο θέμα που δεν αναφέρθηκε είναι οι κρατικέ ενισχύσει. Μεγάλο πρόγραμμα για πολλέ οργανώσει ιδιαίτερα μικρέ, Παρακαλώ τον κύριο Μίτσελ να το σχολιάσει. Οι κανόνε για τι κρατικέ ενισχύσει δηλαδή για τις μικρές οργανώσεις, τι ισχύει. Και το τελευταίο, η απλούστευση για τις αιτήσει. Στις αιτήσει, τεράστιο πρόβλημα. Εμείς εδώ στην Επιτροπή ασχολούμαστε με την απλούστευση των κανόνων να γίνουν πιο εύκολο για λόγους ελέγχου. Θα έπρεπε όμω να ασχοληθούμε και για την απλούστευση κανόνων για τις αιτήσει, για αυτούς που κάνουν αιτήσει, τους αιτούντες. Το παραέχουμε συζητήσει το θέμα. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να μπούμε σε λεπτομέρειες με ανθρώπους που στην πράξη δουλεύουν με τα θέματα αυτά, αυτούς που κάνουν τις αιτήσει, να ξέρουμε τι προβλήματα συγκεκριμένα αντιμετωπίζουν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Παρακαλώ καταρχήν τον κύριο Επίτροπο να απαντήσει και μετά ο κύριος Μίτσελ. ο κύριος Λεβαντόφσκι στα αγγλικά. Γι' αυτό είναι χρήσιμη η ακρόαση, γιατί θα το τι λέει ο κόσμος. Ακούσαμε λοιπόν πολλά σχόλια και για πρακτικές τροπολογίες που δεν χρειάζονται επαναστατικούς κανόνες και αλλαγέ στο δημοσιονομικό κανονισμό. Παραδείγματος καλή πρόσβαση στην πληροφορία. Βέβαια δεν έχει άμεση σχέση αυτό με το δημοσιονομικό προπολογισμό, αλλά κάτι μας δείχνει πώς θα συγχρονιστούν τομεακοί κανόνες. Το ανάφερε και ο κύριος Ματήλα και η κυρία Τότ και η Ίγκε Γκρέσλε. Με την ερώτηση τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορώ να σας αναφέρω τις λεπτομέρειες, να σας αποκαλύψω λεπτομέρειες τι συζητάμε στην Κομισιόν, αλλά επέμενα σε δύο σημεία με πρακτικές ρυθμίσεις. Το ένα είναι η προχρηματοδότηση και πώς γίνεται η ακαθάριση, το clearance. Ένα γνωστό πρόβλημα στο κοινοβούλιο αυτό και στο ηλεκτρικό συνέδριο. Και το δεύτερο, ο συγχρονισμός και η ομοιομορφία κανόνων κατά τομέα με το πνεύμα και το γράμμα του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεν είναι εύκολο αυτό. Κάναμε ένα τεστ σε κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κύριο Ματήλα, την έρευνα. Μακριά διαδικασία συνεργασίας με τον Επίτροπο Γκάγκαν Κουίν που είναι υπεύθυνο για τα θέματα αυτά και η ανακοίνωση της Επιτρόπου ήταν η υπαριθμόν ένα ανακοίνωση και δεν είναι τυχαίο αυτό πριν από το δημοσιονομικό κανονισμό την ανακοίνωση Υπάρχουν ειδικοί δικαιούχοι στην έρευνα και πιστεύω ότι αποδώσαμε ιδιαίτερη προσοχή και είχαμε καλή συνεργασία με την κυρία Γκέγγεν Κουίν για να συγχρονίσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Το ενδιαφέρον για μένα και με ενδιαφέρον άκουσα ο κύριος Μίτσελ να λέει ότι η κρίση κάνει πιο ελκυστική την πολιτική συνοχής καλό σημάδι αυτό για τους μελλοντικού προπολογισμού της Ένωσης και η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ιδιαίτερα σημαντική στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Επίσης η κυρία Τότ αναφέρθηκε σε, σε κάτι που ακούστηκε μάλλον κάτι σαν συντηρητικό σε σχέση με τη δική μας βούληση για επαναστατικές αλλαγές στην προσέγγιση μέσω κόστους κλπ. Και η Concord ακολουθεί μια κλασική προσέγγιση. Το πραγματικό κόστος, το τρέχον κόστος. Εμείς απλώς ανοίγουμε την πόρτα. Το καταποκοπή λάμψαν πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Αλλά μπορείτε να θέλετε να παραμείνετε με το κλασικό καθεστώς ή να περάσετε σε ένα καθεστώς το οποίο να είναι προσανατολισμένο να αφορά την απόδοση ή το τελικό προϊόν. Αναφέρθηκε επίση η επιλεξιμότητα ως προς τον ΦΠΑ. Να σας πω τη δική μου εμπειρία από το 2005. Στο μηχανισμό ισοτιμιών. Στο μηχανισμό ισοτιμιών στους ε, εφαρμοστικούς κανόνες, το άρθρο 8 και με βάση το σημερινό δημοσιονομικό κανονισμό δίνει την ε, δυνατότητα στον διατάκτη να εγκρίνει τους, τις τρέχουσες ισοτιμίες. Όσοι έχουν σήμερα οι χρηματαγορές είναι ιδιαίτερα σημαντικό η απόφαση του διατάκτη σε ένα δύσκολο περιβάλλον στις σχέσεις Ευρωζώνης με την εκτός της Ευρωζώνης δεν θέλω βέβαια να μπω τώρα στο, στο μέλλον της Ευρωζώνης και πώς μπορεί να βελτιωθεί πάντως οι τρέχουσες ισοτιμίες επιτρέπονται ακόμα και με τον σημερινό δημοσιονομικό κανονισμό. Μπορώ γενικά να σας πω ότι εξαρτάται από εσά. Έχει γίνει πρόταση συνεργασία με πολλούς επιτρόπους για τους κανόνες κατά τομέα, όπως σας είπαμε, τη Στάναφο Γκάγκαν για την έρευνα. Τώρα ξεκινάει η φυσιολογική διαδικασία συναπόφασης. Εσείς είστε εκλεγμένοι από το λαό, είστε υπόλογοι στο λαό, στους λαούς, το Ευρωκοινοβούλιο εννοώ. Εγώ το μόνο που μπορώ να υπογραμμίσω είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι τον Ιανουάριο του 2011 του 2012 συγγνώμη και για τη στρατηγική 2020 αλλά και για να έχουμε μια σταθερή βάση εφαρμογής των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτά ήταν τα σύντομα σχόλιά μου. Στα σχόλιά σας πάνω στα προηγούμενα σχόλιά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Μίτσελ. Παρακαλώ να απαντήσετε στην ερώτηση και σύντομα παρακαλώ, το λέω και το εννοώ. Θα σας διακόψω, εάν με κρηγορήσετε. Ναι, φυσικά θα κάνω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ πολύ και για τις ε, δύο ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω ε, τις απαντήσεις. Ε, από την προοπτική των μη κυβερνητικών οργανώσεων, το πιο σημαντικό είναι η ικανότητα να έχει διάλογο με έναν χρηματοδότη, έναν διάλογο ανάμεσα σε δύο φορείς που θέλουν ε, να πετύχει το πρόγραμμα, ε, να μην υπάρχει δυσπιστία ανάμεσα στον ε, χρηματοδότη και στον ετούντα. Κάποια σημεία που θέλω να αναφέρω. Το θέμα της καινοτομία για τον τομέα μας είναι πολύ σημαντικό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή τα χρήματα του Κοινωνικού Ταμείου χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθούν πολιτικές της κυβέρνησης αντί να επιτρέπουν περιθώριο για την καινοτομία και την δημιουργικότητα. Είναι ε, δεξιότητες αυτές ε, που έχουν χαθεί από τον τομέα μας ε, λόγω του μηχανισμού χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ πολύ ότι η αξία των μεγάλων συμβάσεων ε, μειώνουν ε, την, ε, το διοικητικό άχθος, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρές οργανώσεις, τις μικρές κοινότητες να συμμετέχουν στην διαδικασία βελτίωσης της ζωής των πελατών τους με χρήση ευρωπαϊκών πόρων. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, Συμφωνώ να υπάρξει απλοποίηση. Υπάρχει όμως και ανάγκη κατανόησης της ε, κρατικής ενίσχυσης από τις μικρομεσαίες οργανώσεις, ε, από τους μικρομεσαίους φορείς. εάν, ε, υπάρχουν, εάν ο χρηματοδότη είναι ένα συνάδελφος που θέλει να βοηθήσει να πετύχει το πρόγραμμα αντί να είναι κάποιος ε, απόμακρος ε, χρηματοδότης, αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο. Θα είναι χρήσιμο να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ποια είναι η αξία του προγράμματο για την κοινότητα. Όσον αφορά την απλοποίηση ως φορέας λαμβάνουμε ε, χρήματα ε, από εθνικές και από ευρωπαϊκές πηγές. Ε, οι απαιτήσει όσον αφορά το λογιστικό έλεγχο είναι κάπως διαφορετικές. Ένα παράδειγμα. Το διάστημα που πρέπει να διατηρηθούν τα έγγραφα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για το Ηνωμένο Βασιλείο είναι μέχρι το 2025. Ε, για το Progress είναι πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση. Το που θα είμαι εγώ ε, το 2025 δεν το ξέρω, αλλά η οργάνωσή μου έχει την υποχρέωση να διατηρήσει τα έγγραφα αυτά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα ήταν ε, σημαντικό βήμα εάν, ε, ο περιορισμός, εάν το χρονικό διάστημα διατήρησης των εγγράφων περιοριστεί από τα 12 στα 5 ή 7 χρόνια. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο διότι, λόγω του περιορισμένου χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, όσον αφορά τον ε, κύκλο, το, τον κύριο ερωτήσεων και απαντήσεων. Η κυρία Τότα, πολύ λίγο όμως. Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι πολύ σύντομη κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να απαντήσω. Πρέπει να υπερασπιστώ τις θέσεις μου. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον διάλογο που έχουμε με τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια μαζί τους. Επίσης γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο να αλλάξει οποιοδήποτε κανόνα έστω και κατά ένα εκατοστό προς την κατεύθυνση των ε, ε, ε, αποδεκτών. Γι' αυτό δεν υπερασπιζόμαστε μόνο το κλασικό μας καθεστώς, προσπαθούμε να είμαστε και ρεαλιστές. Ειλικρινά, εάν εγώ ήξερα ότι αυτό θα αποτελέσει βάση για τις επόμενες δημοσιονομικές πρόπτικες, δηλαδή αν μιλάμε για τριετίες και έχουμε τώρα μια μεταβατική περίοδο και τότε πραγματικά θα πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες για τις ε, νέες δημοσιονομικές πρόπτικες, διότι τότε θα δραστηριοποιείται το ΙΕΣ, οι ε, αντιπροσωπείες ε, θα δουλεύουν επί τόπου, οι αλλαγές ε, ε, θα ε, αλλάζουν οι κανόνες. Αν το ήξερα αυτό θα είχαμε υποβάλει πολύ πιο ρίζικες προτάσεις. Θα αγράψουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε το έγγραφο αυτό, το οποίο λάβαμε σήμερα μόλις, για από ό,τι φαίνεται υιοθετήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία μέχρι την ηρωστικοποίηση και υιοθέτηση του κανονισμού το 2011. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πράγματι Το Κοινοβούλιο θέλει να διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στην Κομισιόν και στις μη οργανώσεις. Ε, θα ε, δώσω τώρα την προεδρία της ε, σημερινής μας συζήτησης στον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σε αυτή τη φάση ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό εμείς ως συνομοθέτες να ακούσουμε την άποψή σας εμπειρογνωμόνων για να δούμε που υπάρχουν ασθενή σημεία που γίνεται κριτική αλλά μας ε, προτείνεται και βελτιώσεις σε αυτή την νομοθετική φάση χρήσιμες. Και τώρα το λόγο στο Richard Doherty της Deloitte Consulting που θα μας μιλήσει για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού της Ένωσης εμπειρίες από τις τελευταίες αναθεωρήσεις από το 2005 και μετά. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα να μιλήσω σήμερα. Ακολουθούμε το θέμα αυτό. Ως σύμβουλοι και ελεγκτές για πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε στενά με την ε, Κομισιόν σε σχέση με την δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο και επίσης διενεργούμε πολλές ε, έρευνες για αυτές τις δύο επιτροπές ήδη από το 2006. Θα πρέπει να πω ότι ε, πολύ από το υλικό που προετοιμάσαμε έχει ήδη συζητηθεί από τον Επίτροπο και από άλλους ομιλητές. Έχει καλυφθεί. Θα πω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις λοιπόν και στη συνέχεια θα επικεντρωθώ στο τελευταίο τμήμα της παρουσίασής μου αντί να αναφερθώ και πάλι στις επιχορηγήσεις θέματα που ήδη συζητήθηκαν. Νομίζω ότι είναι εύκολο να ασκεί κανείς κριτική σε αυτό το τομέα γιατί αυτοί που εποφελούνται από τον προπολογισμό της ε, κοινότητας ε, και συχνά αυτό είναι πολύ θεμητό ε, επισημαίνουν κάποιες αδυναμίες στη λειτουργικότητα αυτής της διαδικασίας. Και νομίζω ότι αυτό που αυτή η συζήτηση και άλλες συζητήσεις στο πλαίσιο αυτό δείχνουν είναι ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και ότι οι ενδιαφερόμενοι όμως... Α, συγγνώμη, υπάρχει μια βαθμία ορίμανση και οι ενδιαφερόμενοι ε, καταλαβαίνουν τη λογική αυτή της ε, διαδικασίας. Και το έργο των ε, συναδέλφων της Επιτροπής αναγνωρίζεται σε σχέση ακριβώς με το ανοιχτό πνεύμα που επιδεικνύει όσον αφορά την προσέγγιση αυτού του σύνθετου προβλήματος Τη μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού κανονισμού. Όταν μιλάω για περιορισμούς ή καταναγκασμούς θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ένα θέμα ε, ε, όσον αφορά ε, το περιβάλλον διαχείριση στην Επιτροπή σε σχέση με τη ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων μετά από πολλά χρόνια κάποιος ε, συνάδελφος μου είπε ότι χρειαζόμαστε 20 χρόνια για μια τέτοια μεταρρύθμιση. Ίσως αυτό είναι μια υπερβολή, αλλά πραγματικά μας δείχνει πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες όσον αφορά την αλλαγή μιας ε, κουλτούρας ε, διαχείρισης δίκης στην Επιτροπή. πολύ συχνά οι κριτικές έχουν απλουστευτικό χαρακτήρα, κριτικές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους πολιτικούς και όχι αναγκαία από αυτή την κριτική στο επίπεδο των χωρών μελών, ίσως πολύ παραπάνω, που όταν αντιμετωπίζουν κάποιο περιστατικό παρατυπίες και λοιπά διοικητικού τύπου και συχνά με την υποστήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης που είναι άκρητα ε, αμαυρώνουν την εικόνα της Επιτροπής και αυτό δημιουργεί ένα μηχανισμό φυσικής άμυνας, υπερβολική άμυνα, άμυνας εκ μέρους της Επιτροπής. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ισορροπία ε, μεταξύ του θεμητού αιτήματο των ε, αποδεκτών ή δικαιούχων των κοινοτικών κονδυλίων και αυτού του περιβάλλοντος ε, διαχείρισης του, του, του, ήθους, του διαχειριστικού ήθους της Κομισιόν αλλά και της αντίδρασης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όλο αυτό στο πλαίσιο αυτής της ακρόασης προσπαθώντας να πετύχουμε ε, ένα πιο όριμο σύστημα. Όσον αφορά τα σχόλιά μου, θα αναφερθώ στους στόχους της μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού κανονισμού τελευταία πέντε έτη. Θα σχολιάσω τα αποτελέσματα και στη συνέχεια θα υποδείξω ορισμένε ιδέες για το μέλλον. Όπως είπα προηγουμένως, μπορούμε να διατρέξουμε ε, εντάχει τα πρώτα σημεία γιατί νομίζω ότι καλύφθηκαν ήδη. Εν συντομία θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την πλευρά των, ε, της προμήθειας, η Επιτροπή ζητά στις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση να αυξηθούν τα κατόφλια για τις ε, προμήθειες ε, χαμηλού ύψους, προσπαθώντας να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης απόφασης στους διαγωνισμούς στο πνεύμα της νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες, ώστε να αυξηθεί η ποιότητα των προμηθειών μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού. Επίσης να υπάρξει μια ευθυγράμμιση της δικασίας αυτής προποφώντας περισσότερες συμβάσεις πλαίσια και διευκολύνοντα τη σύναψη συμβάσεων και νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε αυτήν την τάση να επικρατεί σε όλα τα θεσμικά όργανα τη κοινότητα που είναι σε θέση να αποφεληθούν αυτέ τι συμβάσει πλαίσια που ξεκινάει η Επιτροπή. Ε, επίσης, όσον αφορά τις τραπεζικές εγγύησεις, που ήταν μια μείζον δαπάνη για τους ενδιαφερόμενους στο παρελθόν. Νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει λυθεί χωρίς αυτονομίωση του δημοσιονομικού ελέγχου. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ο στόχος είναι να απλουστευτούν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με την απλούστευση των αποφάσεων με ψηλότερα κατόφλια για το μοντέλο των καταποκοπήν ποσών, κάτι που είναι ελκυστικό για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ακούσαμε κάποια πράγματα σχετικά σήμερα. Επίσης όλη η, κίνηση, η τάση προς, τα, προς τους ενιαίους συντελεστές, τους τομείς αυτούς και μεγαλύτερη διάρκεια για την υποβολή αιτήσεων, προσφορών ούτως ώστε οι να καταλαβαίνουν τι ακριβώς τους ζητείτε και να προετοιμάζουν τις αιτήσει τους, τις υποβολές προσφορών ε, πιο σωστά χωρίς να αντιμετωπίζουν ε, τις διοικητικές ε, γραφειοκρατικές προκλήσεις που δυσχεραίνουν το έργο τους. Επίσης το θέμα της αυτόματης προχρηματοδότησης και τις μεταρρυθμίσεις για τα επιτόκια που έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα από το συνάδελφο από την πλευρά της έρευνας. Ένας τρίτος τομέας ε, όπου οι μεταρρυθμίσεις ήθελαν να πετύχουν κάποιες αλλαγές ε, αφορούν τη διαφάνεια, δηλαδή μεγαλύτερη σαφήνεια εν σχέση με ποιοι διαφερόμενοι έλαβαν επιχορηγήσεις, ε, καλύτερο feedback για τους μη επιτυχώντες τούντες Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν βελτιώσει από τι υπηρεσίε τη Επιτροπή όσον αφορά ακριβώ αυτό το feedback, ιδιαίτερα την πλευρά των προμηθευτών. Κάτι που είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Και όσον αφορά την πλευρά των επιχορηγήσεων, υπάρχουν ακριβέστεροι ορισμοί, μεγαλύτερη σαφήνεια, περισσότερες ε, πληροφορίες, καλύτερη δημοσίευση και όλα αυτά βοηθούν τους ατετούντες να κατανοούν ε, ε, τι ακριβώς του ζητείτε. Τέλος, όσον αφορά την διαφάνεια, έχουμε από τους ίδιους εξωματογούς της Επιτροπής βοήθημα εργαλεία, όπως είναι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, για τους ε, δυνάμει υποφελούμενους ε, δικαιούχους και μεγαλύτερη σαφήνεια και προστασία. Αυτή είναι η στόχη. Τώρα, όσον αφορά με την δική μας ερμηνεία του τι έχει επιτευχθεί, θα θέλαμε να θέσουμε τέσσερις ή πέντε ορίς, ε, τομείς όπου έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Καταρχήν όσον αφορά ταχύτητα των πληρωμών. Αυτό ήταν ένα σημαντικό θέμα τα τελευταία χρόνια, αλλά ξεκάθαρα θα πρέπει να πούμε ότι καρποφόρησαν οι προσπάθειες και αν και βεβαίω η κατάσταση δεν είναι ιδεώδη, υπήρξε μια σημαντική επιτάχυνση στι διαδικασίε. Όσον αφορά τώρα τη δημοσιονομική ενημέρωση για του ενδιαφερόμενους εν γέννη, η Επιτροπή δημοσιεύει τα δεδομένα για όλου του ενεχόμενου, το Κοινοβούλιο, τι χώρε μέλη, του εξωτερικού οργανισμού κλπ, ούτω ώστε να έχουν μεγαλύτερη εποπτεία στην ε, δημοσιονομική του ε, θέση. Τώρα όσον αφορά τι. Ε, προμήθειες. Οι στόχοι εδώ, όπως σας είπα, έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Μιλάμε για τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού μέσω μιας διαδικασίας δύο σταδίων. Και πολλές υπηρεσίες της Επιτροπής ζητούν μόνο όσους έχουν κερδίσει έναν, μια τέτοια διαδικασία υποβολής προσφορών να εκπληρώσουν όλα αυτά τα κριτήρια. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις υπηρεσίες σε πολλές περιπτώσεις όλοι οι διαγωνισμοί ε, αναγκάζονται να υποβάλουν λεπτομεριακούς φακέλους. Παρ' όλα αυτά έχει επιτευχθεί μια πρόοδο σε αυτό το τομέα. Όσον αφορά τις επιχορήγεις υπάρχει μια μείωση του ε, διοικητικού γραφειοκρατικού άχθους, υπάρχει μια πρόοδο κλπ. Τώρα όσον αφορά τις προκαταχωρήσεις και την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και πάλι θα πρέπει να πούμε ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο απέχει από μια, από μια ιδεώδη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, οι ευρωπαϊκέ υπηρεσίε αρχίζουν να είναι πιο ανοιχτέ ε, προς αυτή την ε, οργάνωση καταχώρηση, προκαταχώρησης των νομικών, δημοσιονομικών στοιχείων των ενδιαφερόμενων κλπ. Τώρα, όσον αφορά την αρνητική πλευρά, δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα όσα είπαν ήδη συνάδελφοι με όρους ε, δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όσον αφορά το διοικητικό άχθος ε, διάφορες ασυνέπειες που υπάρχουν όσον αφορά την αρμηνία και εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων. Βεβαίω ε, ε, χιλιάδες αξιωματούχοι της Κομισιόν προσπαθούν να διχριστούν τη διαδικασία, αλλά αν ο βαθμός σύγχυσης και διοικητικού άχθους είναι τέτοιος που τελικά οδηγεί, τελικά γίνεται αντικίνητρο για τη συμμετοχή, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες από την πλευρά της Επιτροπής. και μάλιστα έγινε σχετικά μια ειδική ακρόαση ε, για τα ερευνητικά προγράμματα συγκεκριμένα. Τέλος, για να επανέλθω στα όσα είπα για την κουλτούρα που επικρατεί, τα ήθη της Κομισιόν. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα συνεχής φόβος ε, έναντι ε, σφαλμάτων και μία έρευνα που έγινε πριν από μερικά χρόνια εξέταζε το θέμα της εξοπιστίας των αξιωματούχων και δεν ήταν τόσο πολύ ο κίνδυνος νομικής φύσεως που αντιμετώπιζαν, αλλά ένας πιο φυσικός φόβος, συνθισμένος φόβος που έχει κάποιος που δεν θέλει να ε, αντιμετωπίσει σαν κάποιος που έχει διαπράξει ένα σφάλμα. Και ε, στη συνέχεια προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε ε, το βαθμό εμπιστοσύνης των αξιωματούχων, των υπαλλήλων της Επιτροπής όσον αφορά αυτό το ενδεχόμενο ενό σφάλματος, ούτως να αυξηθεί και η αποτελεσματικότητα η αποτελεσματικότητα στο διαχειριστικό του ρόλο για να υπάρξει σωστή εφαρμογή των κανόνων. Τώρα, και εξετάζω στο μέλλον. Όσον αφορά την πλευρά τη διαδικασία, εδώ επέλεξα πέντε σημεία τα οποία πιστεύω είναι αντιπροσωπευτικά για αυτό το οποίο συζητούμε και που θα μπορούσε να βοηθήσει. Ο βαθμός αποδεκτού σφάλματος, ε, εδώ βλέπουμε ότι τα πράγματα εδώ κινούνται ξεκάθαρα και αυτά είναι πολύ καλά νέα. Οι κανόνες για την ε, κοινοποίηση όσον αφορά τα ήθη της Επιτροπής, η βελτίωση αυτού του ε, περιβάλλοντος, γιατί υπήρξαν ε, περιπτώσεις όπου όλο και περισσότερο πάλι της Επιτροπής ενέχονται στη διαδικασία βελτίωσης των, ε, της κατάστασης και των διαδικασιών. Και νομίζω ότι με αυτό μπορεί να επιτευχθεί πράγματι μια πρόοδος και επιτάχυνση των διαδικασιών όσον αφορά την ανακοίνωση ξεκάθαρων κατευθυντήριων γραμμών και σε σχέση με τον έλεγχο τέλος και αυτό φάνηκε στην ακρόαση για την χρηματοδότηση της έρευνας. Εδώ βλέπουμε μία πρόοδος όσον αφορά το περιθώριο αποδεκτού σφάλματος και νομίζω το μέλο του ελεγκτικού συνεδρίου που θα λάβει το λόγο αργότερα θα το, αναλα... θα το αναφέρει. Αλλά η πρόληψη των σφαλμάτων και η διασφάλιση να μην ανακύψουν τα σφάλματα πολύ περισσότερο παρά η επιβολή κυρώσεων νομίζουμε ότι είναι ενδεγμένος τρόπος για να κινηθούμε. Και τέλος μια ε, τελευταία διαφάνεια που διευρύνει το φάσμα ως προς την εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων. Ο δημοσιονομικός κανονισμός περιλαμβάνει το άρθρο 27.3 που λέει ξεκάθαρα ότι όλες οι δραστηριότητες στην Επιτροπή θα πρέπει να πλαισιώνονται ε, από ξεκάθαρους στόχους που θα πρέπει να προσμετρώνται από δείκτες αποδοτικότητας και θα πρέπει να υπάρχει σχετική αναφορά, η παρακολούθηση και η λογοδοσία. Και οι αρχές αυτές μέχρι στιγμής δεν έχουν εφαρμοστεί στη μεθοδολογία της ε, Κομισιόν με το πνεύμα αυτό. Και η διαφάνεια αυτή δείχνει ορισμένους από τους δείκτες της ε, σωστής αποδοτικότητας. Το ήθος ακριβώς της, ε, του ετήσιου προγραμματισμού σε κάθε γενική διεύθυνση και της, του ετήσιου reporting εν σχέση με το πώς επιτυχάνονται αυτά τα προγράμματα. Αυτό το ήθος έχει φτάσει στην αρχική φάση ορίμανσης. Βεβαίως ε, δεν έχουμε μέχρι στιγμής φτάσει στο επίπεδο του στρατηγικού προγραμματισμού στο οποίο στοχεύουμε. Και νομίζουμε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι ιδιαίτερε αποφαλέ για την Κομισιόν, ούτε ώστε να υπάρξει μια μεγαλύτερη σαφήνεια εν σχέση με την ανάπτυξη των πόρων και την ε, δημιουργία μιας ουσιαστικής αξιολόγησης που θα επιτρέπει ε, στην Κομισιόν να προγραμματίζει πιο αποτελεσματικά όχι μόνο σε αιτήσια βάση αλλά βάση ακριβώς της λογικής του πολιετούς προγραμματισμού για τον προγραμματισμό των ε, δραστηριοτήτων της ε, Κομισιόν, ούτως ώστε να υπάρχει μια συνεπής καθοδήγηση όχι μόνο της λειτουργίας της ίδιας Επιτροπής, αλλά και των άλλων θεσμικών οργάνων και της αρχής του προπολογισμού, τους ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις επί των πραγματικών δεδομένων. <coughs> Ευχαριστούμε. Και το λόγο στον κύριο Ντομένικο Ντιμαρτίνο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις υποχρεώσεις των κρατομενών στην εκτέλεση του προπολογισμού με βάση το νέο άρθρο 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης. Έχει το λόγο κύριο Ντιμαρτίνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για το ότι μου δώσατε την μεγάλη ευκαιρία να πάρω μέρος στη συνεδρίαση της Επιτροπής σας και επειδή δεν έχουμε χρόνο δεν θα αναφερθώ καθόλου στην εισαγωγή της ε, ομιλίας μας για τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις που καθορίζουν την συνθήκη της Λισαβόνας και την θέση της ισχύ και τα χαρακτηριστικά των κανόνων που αναφέρονται στη συνθήκη. Μιλώντας λοιπόν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών με βάση το άρθρο 317 της συνθήκης, θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα λογικό κριτήριο ερμηνείας σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των κανόνων και με άλλους κανόνες που, ο, της συνθήκης η υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να δώσει μια συγκεκριμένη στάση συνεργασίας με την Κομισιόν για την προετοιμασία του κοινωνικού προϋπολογισμού και την νόμιμη εφαρμογή του. Το άρθρο αυτό απαιτεί και τη συνεργασία των κρατών στην επεξεργασία του προϋπολογισμού και την ευθύνη της Κομισιόν για τη σωστή χρήση των πόρων με βάση τις αρχές μιας καλής οικονομικής διαχείρισης σε σχέση με τους κοινωτικούς στόχους. Η σωστή συνεργασία εκ μέρους των κρατών μέλων με την Κομισιόν θα μετρηθεί και στην, φάση, στην πρώτη φάση των στοιχείων που θα μπουν στον προπολογισμό και στη φάση ελέγχου και εφαρμογής του. Το άρθρο 310 της ηθικής προβλέπει όλα τα έσοδα και δαπάνε τη Ένωση πρέπει να πλούν αντικείμενο πρόβλεψης για κάθε οικονομικό έτος άσκηση να είναι γεγραμμένο στον προπολογισμό με βάση ένα πολιετές πλαίσιο που αναφέρεται σε διάρκεια ποτέ κάτω των πέντε ετών. Επίσης το άρθρο αυτό προβλέπει ο προπολογισμό τα έσοδα και οι δαπάνε πρέπει να είναι ισοσχελισμένα. Υπάρχει δηλαδή η αρχή, όλοι οι ήδη πόροι της Ένωσης θα πρέπει να θεωρούνται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διάρκεια αυτού του έτους μέσω της συνεργασίας αυτής η οποία αναφέρθηκε προηγουμένως με τα κράτη-μέλη. Συνεπώς αυτή η συνεργασία λειτουργικά είναι σημαντικό στοιχείο αναφοράς για την Κομισιόν και σε σχέση με τα κονδύλια που χρειάζονται για να επιτευχθούν οι κοινωτικοί στόχοι και σε σχέση με τη σωστή προγραμματική εφαρμογή της αρχικής πρόβλεψης του προπολογισμού. Η ανάγκη λοιπόν συνεργασίας των κρατών μελών σε σχέση με τα αποτελέσματα που θέλει να πετύχει η Ένωση και σύμφωνα με τις προβλέψεις του προπολογισμού εισάγει την ανάγκη πρόληψης σε σχέση με τα στοιχεία που δίνουν τα κράτη-μέλη πριν συνταχθεί ο προπολογισμό και ενδεχόμενες κυρώσεις σαφείς στη φάση εφαρμογής του προπολογισμού με βάση τη δημοσιονομική πειθαρχία αν τυχόν γίνει παράνομη χρήση των κονδυλίων σε σχέση πάντα με τις προγραμματικές δηλώσεις και προβλέψεις. Συνεπώς είναι υποχρέωση των κρατών μελών να διατυπώνουν στην πρώτη φάση του προπολογισμού σωστές ενδείξεις σχετικά με τις προβλέψεις δαπανών με βάση πραγματικές ανάγκες και προοπτική ασφαλούς και αξιόπιστης εφαρμογής των αποτελεσμάτων προς το συμφέρον και των κρατών μελών και της Ένωσης. Είναι επομένως υποχρέωση των κρατών μελών να εγγυηθούν την εφαρμογή με σεβασμό των κανόνων και των αρχών της Χριστούς, χριστής δημοσιονομικής διαχείρισης των στόχων με αναφορά στους οποίους έγιναν οι προβλέψεις του προπολογισμού που σημαίνει να ανταποκρίνει στην πραγματικότητα στις ανάγκες του κράτους συγκεκριμένων τομέων όσον αφορά προκειμένου να δοθούν τα κονδύλια στα πλαίσια της πρόβλεψης του ετήσιου προπολογισμού. Ειδική λοιπόν υποχρέωση. Όχι γενική συνεργασία όπως ορίζει το άρθρο 317 προκειμένου να υπάρχει μια σωστή παροχή συμβολής όπως απαιτεί ο προπολογισμό, απορρέει η ανάγκη άλλου κανόνα που την προβλέπει η συνθήκη, το άρθρο 122, που ρυθμίζει τις σχέσεις οικονομικής πολιτικής. Αν υπάρχει ε, διαφωνία μεταξύ αυτού που λέει η Κομισιόν και των μέτρων που ενέκρινε ένα κράτος, μπορεί να οριστούν εκεί μέτρα πολυμερούς εποπτείας. Στην περίπτωση που η Κομισιόν θεωρήσει ότι δεν συμφωνεί με το κοινοτικό δίκαιο τα μέτρα ενός κράτους μέλους, προβλέπεται η δυνατότητα προειδοποίησης στο κράτος μέλος και ενδεχομένως θα δημοσιευθούν οι συστάσεις αυτές. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εγκριθούν μέτρα που προβλέπει η διαδικασία πολυμερούς επιτήρησης. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τέτοιου είδους προβλέψεις πειθαρχικού χαρακτήρα με τον ίδιο στόχο που είναι κοινό είτε για την Ένωση είτε για τα κράτη-μέλη είναι αναγκαίο αναγκαίος ο μέγιστος σεβασμός εκ μέρους των κρατών μελών των υποχρεώσεων που έχουν για τη συνεργασία όπως προβλέπει το άρθρο 317 της Συνθήκης. Αυτό είτε γενικά σε σχέση με τα αποτελέσματα της ετήσιας άσκησης ή και πολυ, πολυετούς φυσικά στις προβλέψεις του προπολογισμού είτε ειδικά σε σχέση με την καταπολέμηση της απάτης που προβλέπει το άρθρο 310 της συνθήκης και ρητά όπως εκφράζεται στο άρθρο 325. Η πρόσβαση σε παράνομες δραστηριότητες συγκεκριμενοποιείται όσον αφορά την προστασία της νομιμότητας στον έλεγχο του κατά πώς εκτελούνται οι δραστηριότητες στα κράτη-μέλη και με τη μέγιστη απέτηση συνεργασίας από τα κράτη-μέλη προκειμένου να έχουμε θετικά αποτελέσματα σε θέματα καταπολέμησης της απάτης εκ μέρους της Ένωσης. Ανεξάρτητα από την ε, ανάλυση των μορφών παρανομίας, ένας ανάλογος κίνδυνος κακής χρήσης των κονδυλίων και όχι σαφή παροχή πληροφοριών για να καθοριστεί ο προπολογισμό. Πρέπει να αφορά όλες τις πρωτοβουλίες που δεν έχουν στόχο αποτελέσματα συλλογικού συμφέροντος γιατί το συλλογικό συμφέρον θα πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας που θα καθορίζει την προοπτική και τους στόχους και για τους πολίτες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη επιπλέον προβλέπει τα μέτρα εθνικού χαρακτήρα των κρατών μελών με βάση τις αρμοδιότητες που υπάρχουν προκειμένου να καταπολεμηθεί, καταπολεμηθούν οι απάτες στο βαθμό που τα κράτη-μέλη καλούνται να εγκρίνουν μέτρα έτσι ώστε η απάτη να μην γίνεται σε βάρος του κοινού συμφέροντος. Σε περίπτωση πρωτοβουλειών που χρηματοδοτούνται από κοινωτικές οργανώσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη υπ' αυτή την έννοια καλούνται να συνεργάζονται με την Κομισιόν για να οργανώνει τα μέτρα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων που αποκλείουν μεν δυνατότητα απάτης, ταυτόχρονα καθορίζουν την προσφυγή των αρμόδιων αρχών σε στενή οργανική συνεργασία έτσι ώστε η χρήση των κοινωνικών κονδυλίων να συντονίζεται με τους στόχους που είχαν οριστεί εξ αρχής. Έτσι πρέπει να ερμηνεύσουμε το άρθρο 17 της συνθήκης το οποίο ορίζει το ρόλο και την ευθύνη των κρατών μελών πιο ευρύ από μια απλή γενικού χαρακτήρα συνεργασία. Ο όρος συνεργασία στο άρθρο 317 ορίζει και την και ευθύνη του κάθε μέρους δηλαδή η υποχρεωτική δραστηριότητα ελέγχου και λογιστικής αναθεώρησης για τα κράτη-μέλη στην εκτέλεση του προϋπολογισμού προβλέπει το πώς κάθε όργανο θα πρέπει συμμετέχει στην, στο πώς διαχειρίζεται τις δαπάνες του Βέβαια, αυτό είναι ένα κριτήριο αλληλεξάρτησης μεταξύ της ευθύνης και της δραστηριότητας συνεργασίας μεταξύ των κρατομελών αφενός και της Κομισιόν αφετέρου. Και υπάρχει δυνατότητα άσκησης με ένα είδος αυτοπροστασίας στην εφαρμογή του προπολογισμού όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των στοιχείων που δίνουν τα κράτη-μέλη και την αίσθηση ότι αυτά τα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες υπάρχει λοιπόν μια μορφή αυτοπροστασίας με τη δυνατότητα που έχει η Κομισιόν να περάσει κονδύλια από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, από γραμμή σε γραμμή του προπολογισμού. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα να καταγγελθεί η μη τήρηση εκ μέρους των κρατών μελών του κριτηρίου χρηστής συνεργασίας όταν υπήρξε ένα αίτημα εκ μέρους της Κομισιόν για διευκρίνηση και να έχει δημοσιευτεί μάλιστα όταν το κράτος μέλος επιμένει στη συμπεριφορά του να μην τηρεί την ομοθεσία ή η αιτιολόγηση που έδωσε δεν οδηγεί ουσιαστικά στο να δικαιολογεί τα μέτρα αυτά, δηλαδή ότι δεν τα δέχεται η Κομισιόν, τότε η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία παράβασης όπου να αμφισβητήσει τα μέτρα αυτά και στην πρώτη αυτή φάση αμφισβήτησης δίνεται η δυνατότητα στην Κομισιόν αν τυπικά και ουσιαστικά το κράτος μέλος δεν τηρεί το άθρο 317 μπορεί η Κομισιόν να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ληφθούν μέτρα. Έτσι θα πρέπει να δούμε το πραγματικό περιεχόμενο του άρθρου 317 και όχι με την προσφυγή σε ένα ερμηνευτικό κριτήριο μόνο κατά γράμμα, να το δούμε στην πράξη σε σχέση το περιεχόμενό του με τα υπόλοιπο κομμάτι της συνθήκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Δημαρτίνο, Μαρτίνο. Επόμενος συζητητής, ο αντιπρόεδρος του Γερμανικού Ελεκτικού Συνεδρίου, Νόρμπερτ Χάουζερ, για τη δήλωση αξιοπιστίας των ομοσπονδιακών συστημάτων στο πλαίσιο της επεμβλημένη διαχείρισης με βάση το άρθρο 53β του Δημοσιονομικού Κανονισμού της Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που θα έχω τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω κάποιες παλιές και νέες σκέψεις θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει ως εξή, λέγοντας ότι η Ευρώπη έχει ένα πρόβλημα. Μετά το 1994 ε, εξεπλάγημεν, αργότερα πια όμως ε, δεν ε, μας εξέπλητε, ε, το ότι είχαμε πολλές δηλώσεις αξιοπιστίας. Αργότερα ακούστηκε ότι οι πόροι δεν ε, χορηγούνταν σωστά και ότι το περιθώριο λάθους ε, ανερχόταν σε 11%. Αυτό ε, δυσαρεστεί και εσάς ως βουλευτές και την Κομισιόν, ελπίζουμε, και αυτό δυσαρεστεί και τους φορολογούμενους ε, που πληρώνουν. Και αναρωτιέται κανείς τι γίνεται λοιπόν με αυτό. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Κάθε χρόνο λαμβάνεται την πληροφορία ότι δεν λειτουργεί το σύστημα, το ε, περιθώριο λάθους παραμένει μεγάλο, ναι με κάποιες μικρές αποκλήσεις, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Έτσι λοιπόν, ακούστηκε η ιδέα, ας έχουμε μια ετήσια σύνοψη. Αυτά που προβλέπονται στους τομεακούς κανόνες, ε, κάθε φορέας υποβάλλει αυτά που πρέπει, κοιτάμε τι έχουμε ε, συλλέξει και ε, προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε αυτά, ε, να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Στην Γερμανία, που είναι ομοσπονδιακό κράτο, τα 16 κρατήδια υποβάλλουν έγγραφα και υπάρχει κάποιο που τα συνθέτει αυτά και τα στέλνει στην Ευρώπη. Ως, εξωτερική, ως εξωτερικός λογιστικός έλεγχος έχουμε σκεφτεί ε, τι ε, επιφέρουν όλα αυτά. Έχει ε, επιφέρει προστιθέμενη αξία, υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα με το σύστημα αυτό, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως όχι. Αν σκεφτεί κανείς σε ποιο οικονομικό ε, ε, έτος αναφέρεται η συνθετική έκθεση ε, και η δήλωση αξιοπιστίας του ελεγκτικού συνεδρίου, θα δείτε ότι υπάρχει ένα κενό, διότι η δήλωση αξιοπιστία του ελεγκτικού συνεδρίου αναφέρεται στο έτος νήμιον 1, ενώ η συνθετική έκθεση αναφέρεται στο νήμιον 2. Δηλαδή, αν βρισκόμαστε στο 2010, το στο 2009 αναφέρεται η δήλωση αξιοπιστία, ενώ η συνθετική έκθεση αναφέρεται στο 2008. Τι κερδίζουμε λοιπόν, τίποτα. Διαφροντικά ταμεία. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα κενό 1,5 μήνα. Στην ε, ετήσια συνθετική έκθεση ε, για τα ταμεία αυτά βλέπουμε ότι αναφέρονται μέχρι την 15η ε, Οκτωβρίου κάθε έτους, ενώ η δήλωση εξοπιστίας αναφέρεται στο διάστημα μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Υπάρχει λοιπόν κενό ανάμεσα σε αυτό που θέλει το ελεκτικό συνέδριο και σε αυτά που θα μπορούσε να βοηθήσει εσά. Το ελεκτικό συνέδριο της Αυστρίας κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και έχουν ε, αναθέσει έρευνα στην ΆΙΠΑ και το ερευνητικό αυτό Ινστιτούτο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ετήσια συνθετική έκθεση δεν επιφέρει καμία προστιθέμενη αξία. Τότε σκεφτήκαμε ωραία, ας υποβάλουμε εθνικές δηλώσεις από κάθε κράτος μέλος. Υπάρχουν κάποιες εθνικές δηλώσεις μόνο που δεν είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν και αυτές δεν μας βοηθάνε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένο συμπέρασμα, διότι αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε, και θα επανέλθω σε αυτό, είναι πού έγιναν τα λάθη και γιατί έγιναν τα λάθη. Αυτή η ανάλυση λαθών δεν έχει υποβληθεί ακόμα σε εσά και κανείς δεν την κάνει την ανάλυση λαθών αυτή. Οι ε, εθνικές δηλώσεις λοιπόν δεν μας βοηθούν. Έχουμε λάβει εθνικές δηλώσεις από διάφορα κράτη-μέλη και διαπιστώνουμε ότι δεν είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. Και εκεί λοιπόν δεν μας βοηθάνε καθόλου οι εθνικές δηλώσεις. Εάν θέλετε εθνικές δηλώσεις από τα κράτη-μέλη, τότε θα πρέπει να υπάρχει σαφής νομική βάση, θα πρέπει να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους και αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να υπαγορεύει τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στι εθνικές δηλώσεις, με ποια πρότυπα θα ε, δηλώνεται, πώς θα πρέπει να ε, εκπονούνται, να δομούνται αυτές οι εθνικές ε, δηλώσεις, ώστε κάθε κράτος μέλος να απαντάει στις ίδιες ερωτήσεις, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε τα αποτελέσματα των εθνικών αυτών δηλώσεων. Έτσι θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσατε βέβαια και το αναφέρατε αυτό το πρόβλημα να αναρωτηθείτε τι στοιχίζει ένας τέτοιος λογιστικός έλεγχος. Και θα πρέπει βέβαια ε, το κόστος ε, να ε, είναι αναλογικό προς το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι λοιπόν ποιο θα πρέπει να το ελέγχει αυτό, η Deloitte, το εξωτερικό οικονομικό έλεγχο. Φυσικά ο εξωτερικό λογιστικό έλεγχο είναι διατεθειμένος να εξετάσει τέτοιε εθνικέ δηλώσει. Το μόνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ο εξωτερικός λογιστικός έλεγχος να μην αναλαμβάνει εκτελεστικά ε, καθήκοντα. Αυτή τη στιγμή διότι έτσι δεν θα παρέχεται η ανεξαρτησία η αυτονομία του εξωτερικού ε, ε, λογιστικού ελέγχου και έτσι δεν θα ε, διασφαλίζεται η αντικειμενικότητά του. Δηλαδή θέλουμε ε, εξωτερικό λογιστικό έλεγχο αλλά που να είναι εκτός της τελεστικής διαδικασίας. Όσον αφορά τις δηλώσεις αξιοπιστίας του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αυτό δεν λέει πώς, τι μορφή θα πρέπει να έχει μια τέτοια δήλωση αξιοπιστίας. Αναφέρεται μόνο ότι θα πρέπει να υποβάλλεται ετησίως. Εάν δεν υπάρχει ικανοποίηση με την δήλωση αυτή αξιοπιστίας και άκουσα πολλές επικρίσεις και στην αίθουσα αυτή για το θέμα αυτό, τότε αλλάξτε κάτι έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε πρωτοβουλία και να προχωρήσετε στο θέμα αυτό. Τι θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν. Σήμερα λαμβάνουμε δηλώσεις αξιοπιστίας για όλα τα θέματα. Να το πω χοντρά οι ελιές στην Ελλάδα συγκρίνονται με τις ε, ελιές στη Φιλανδία. Προφανώς δεν θα υπάρχουν ε, ελιές στη Φιλανδία, αλλά το ποσοστό λάθους είναι όμοιο. Γίνεται λοιπόν σύγκριση στο επίπεδο του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα για την αγορά εργασίας, ε, πώς λειτουργούν στον Νότο και πώς λειτουργούν στο Βορρά. Αυτό δεν λειτουργεί. Χρειάζεστε αποτελέσματα ανακράτως μέλος. Θα πρέπει να γνωρίζετε τι περιθώριο λάθους υπάρχει, για ποιο ταμείο, σε ποιο κράτο μέλο. και θα πρέπει να ξέρετε πού οφείλεται αυτό. Τα αποτελέσματα αυτά δεν θα τα λάβετε σήμερα. Το ε, ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι δεν έχουμε αρκετό προσωπικό ε, για κάτι τέτοιο, δεν έχουμε αρκετού ελεγκτές. Φροντίστε λοιπόν να έχει το ελεγκτικό συνέδριο αρκετού ελεγκτέ για να μπορεί να ε, ανταποκριθεί στην απέτηση αυτή. Δηλαδή, δήλωση αξιοπιστία αναχώρα, ανά διαφορετικό ταμείο, ώστε να μπορείτε να κάνετε ανάλυση, να βρείτε πού προέκυψαν τα λάθη αυτά για να μπορέσετε να τα λύσετε. Η Κομισιόν ε, έχει υποβάλει πρόταση σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει το άρθρο 53α στο μέλλον. Έχω μια ερώτηση, διότι λίγο με ενοχλεί το ότι δεν καταλαβαίνω αυτά που διαβάζω. Στο άρθρο 53, παράγραφος 4, ε, αναφέρονται τα bots accredited και στο γάμα C λέει ότι θα υπόκεινται σε εξωτερικό ανεξάρτητο έλεγχο. Η λειτουργία αυτή θα είναι ανεξάρτητη από το credited body, το διαπιστευμένο φορέα. Αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες αυτές υπόκεινται απλά στον έλεγχο, σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχονται. Σημαίνει ότι θα ελέγχονται μία φορά το χρόνο, σημαίνει ότι θα ελέγχονται τακτικά. Σημαίνει ότι θα μπορούν να ελέγχονται σε μη τακτά χρονικά διαστήματα. Ποιος ελέγχει. Ποιος είναι ο ελεκτικός φορέας ο οποίος ε, ε, ενεργεί ανεξάρτητα από το διαπιστευμένο φορέα. Και στο 53-4 γ προκύπτει και εδώ το ερώτημα ποιος κάνει τους εξωτερικούς ελέγχους του αρμόδιου φορέα. Και εδώ το 53α δεν δίνει καμία απάντηση. 53α5 δέλτα. Ποιος θα πρέπει να εκπονεί τη γνωμοδότηση για τη δήλωση αξιοπιστίας. Ε, ποιος θα το υποβάλει αυτό στην Κομισιόν. Θα ήμουν ευγνώμων εάν θα μπορούσαμε να ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα αυτά. Και για να κλείσω τη σύντομη μου παρουσίαση, να σας παρακαλέσω και πάλι, φροντίστε να γίνεται ανάλυση των λαθών, να είναι σαφές πού έχουν γίνει τα λάθη, ποιος έχει κάνει τα λάθη. Όταν έχουμε αυτά τα αποτελέσματα μπροστά μας θα είναι εύκολο να αποφύγουμε τα λάθη ακριβώς όπως ζήτησαν και πρότειναν οι προλαλήσαντες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Χάουγκερ. Χάουζερ και αρχίζει η συζήτηση. Κύριε Γκρέσλε πρώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Και το δεύτερο τμήμα της παρουσίασης ήταν εντυπωσιακό ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ για τον κόπο που κάνατε και την απόδειξη ότι σε δέκα λεπτά μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα. Έχω ορισμένα ερωτήματα. Αυτά τα οποία μας απασχολούν εδώ κυρίως είναι οι παραβιάσεις των χωρών μελών στο ελληνικό παράδειγμα μπορούμε να διαπιστώσουμε πολλά πράγματα. Και τότε έχουμε ένα πρόβλημα με την Ελλάδα. Αυτό ο έλεγχο του προπολογισμού το ήξερε πριν ε, από άλλου. Αυτή είναι η χμή του η κορυφή του παγόβωνου. Όταν εμεί αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα, ξέρουμε τι θα γίνει με του υπολείπου. Η Κομισιόν ε, υπόκειται σε ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων. Το ερώτημα είναι το εξή. Θα πρέπει να υποκινήσουμε την Επιτροπή ούτω ώστε να διώκει αυτόματα τις παραβιάσεις των χωρών χωρίς να προηγείται μια συζήτηση. Βλέπουμε τι γίνεται με το ευρώ και βλέπουμε το τίμημα που πληρώνουμε σχετικά δεν είναι δυνατόν να κάνουμε του ανθρώπου πιο θαραλέου από ό,τι είναι. Αλλά για μας αυτό ε, θα ήταν σημαντική η επισήμανση, η ιδέα του πώς μπορούμε να παρενέσουμε την Επιτροπή αυτόματα να διώκει τις νομικές παραβιάσεις των χωρών. Γιατί κάθε φορά που γίνεται σχετική συζήτηση ε, ε, δεν βρισκόμαστε στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου και τελικά κερδίζει αυτός που είναι ισχυρότερος ή αυτός που δίνει τα περισσότερα χρήματα κλπ. Κάτι που κάνει περίπου η Γερμανία αυτή τη στιγμή και κατευθύνει τα πράγματα. Ε, δεν χρειαζόμαστε λοιπόν μια πιο, ένα πιο ωραίο δημοσιονομικό κανονισμό, πιο εξορισμένο ή με πιο πολλέ λεπτομέρειε, αλλά που δεν εφαρμόζει κανεί. Όχι, να δούμε τι γίνεται με αυτέ τι νομικέ παραβιάσει των χωρών. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο η Επιτροπή μετά την παρέτηση του κυρίου Επιτρόπου ε, είναι ικανή να μιλήσει προς τα έξω. Αλλά νομίζω ότι ε, θα πρέπει να είμαστε ευνόμονες για την επισήμανση των ασαφιών εδώ. Για παράδειγμα η έννοια του αποδεκτού περιθωρίου σφάλματος θα πρέπει να δούμε ότι δεν σημαίνει, ότι αλλαγή δεν σημαίνει ότι είναι μια βελτίωση. Παραμένουν πολλές ασάφειες, πολλές ε, ε, βεβαιότητες και νομίζω ότι είναι αναγκαίο να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σχέση με το θέμα ακριβώ του ανεκτού σφάλματο. Γιατί το άρθρο 28 το οποίο έχει παρουσιαστεί εδώ σα λέω ευθύ εξ αρχή ότι είναι εντελώ ανακριβέ και αόριστο ε, είναι η καυτή πατάτα που μας πετάνε και μας λένε τώρα δείτε εσείς τι θα κάνετε. Δεν είχα φανταστεί έτσι τα πράγματα, όχι. Και έχω και ένα ερώτημα όσον αφορά την ποιότητα των ελεκτικών συνεδρίων. Και εδώ πραγματικά θα ήθελα να ρωτήσω τον Ιταλό εμπειρογνώμονα, ο οποίος ασχολήθηκε με τη συνθήκη του εξή. Όταν πρόκειται για τον εξωτερικό οικονομικό έλεγχο, είναι ένα πραγματικό τσίρκο εδώ. Και πάλι με αυτό εννοώ τους Έλληνες φίλους, ε, και θα ήθελα να πω ότι πριν συμπεριλάβουμε την έννοια του σεβασμού της ανεξαρτησίας, κάτι που κάναμε τους Έλληνες φίλους μας και δεν μας οδήγησε πουθενά, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς ε, γίνεται και πώς μπορούμε να πιέσουμε μια σωστή μεταρρύθμιση των ελεκτικών συνεδρίων, ώστε το ελεκτικό συνέδριο είναι ένα εξάρτητο σώμα το οποίο να δεσμεύει όλους τις ίδιες διεθνείς αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο. Ο Γενικός Διευθυντής Ανζέν. Σε σχέση με το ερώτημα της κυρία Γκρέσλε. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με το τελευταίο σημείο που έθεσε η κυρία Γκρέσλε, όσον αφορά το περιθώριο αποδεκτού σφάλματος. Παράλληλα με την προσαρμογή της ε, πρότασής μας για την αναθεώρηση του κανονισμού έγινε η πρόταση για ένα έγγραφο που αφορά ακριβώς το περιθώριο ανεκτού σφάλματος που έρχεται να συμπληρώσει ή μάλλον να διευκρινίσει τις προτάσεις που έγιναν σε σχέση με το άρθρο 28β και θα ήθελα εδώ ίσως να πω δύο πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά το περθώριο σφάλματος ή το ποσοστό σφαλμάτων μπορεί να υπολογιστεί σε αιτήσια βάση. Και στις περισσότερες περιπτώσεις εργαζόμεθα με προγράμματα που είναι πολυετή προγράμματα και που σε πολλές περιπτώσεις τα σφάλματα τα οποία ανεχνεύονται το, ε, το έτος χ διορθώνονται στο έτος ψ και τα ποσοστά σφάλματος έτσι όπως αναφέρονται στο τέλος των περιόδων είναι κατώτερα από τα ποσοστά σφαλμάτων τα οποία έχουν αναγνωριστεί ε, μια συγκεκριμένη χρονιά. Δεύτερον και ως απάντηση σε αυτό που είπε ο κ. Χάουζερ προηγουμένως θα ήθελα να πω ότι τα πέντε τελευταία έτη όσον αφορά την διαχείριση των χωρών μελών, τα ποσοστά ασφαλμάτων πάνω από το 5% πέρασε από το 60% στο 30%. Έγιναν λοιπόν σημαντικές ε, προσπάθειες και που καρποφόρησαν. Τρίτον, σε σχέση με, τα, με το περιθώριο αποδεκτού σφάλματος, με το αποδεκτό περιθώριο σφάλματος. Όπως είπε ο Επίτροπος προηγουμένως, το ζητούμενο δεν είναι να ικανοποιήσουμε ένα ποσοστό σφαλμάτων, αλλά το ζητούμενο για την Επιτροπή ακριβώς στο πλαίσιο της πρότασής της είναι να συνεχίσει να ασκεί τη μεγαλύτερη δυνατή εποπτεία για να μειώσει και να ε, ενεργοποιήσει όλα τα μέσα για να μειώσει τα περιθώρια σφαλμάτων. Δηλαδή υπάρχει ένα στάδιο μετά από το οποίο το κόστος ελέγχου είναι τόσο μεγάλο που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο από τις οικονομίες που γίνονται μειώνοντας το ποστό των σφαλμάτων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για διαχείριση των δημόσιων χρημάτων των χρημάτων του φορολογούμενου. Δηλαδή το να ξέρουμε σε ποια στιγμή βρισκόμαστε σε μια στιγμή ισορροπίας μεταξύ ακριβώς της αιμονής ελέγχου των δαπανών, του στόχου ε, μείωσης των σφαλμάτων και από την άλλη του κόστους που συνεπάγεται ο λόγο έλεγχος. Εδώ λοιπόν αυτά που θα μπορούσα να πω σε σχέση με την ε, παρέμβαση της κ. Γκρέσλε. Και επίσης θα ήθελα να διορθώσω, αν με επιτρέπετε, ένα σφάλμα στην παρουσίαση του κυρίου Χάουζερ, ο οποίος μας λέει ότι στην πραγματικότητα οι ιδιωτικά ταμεία παρουσιάζουμε την ετήσια σύνοψη του άρθρου ε, του, του έτους ε, νήμιον 2. Όχι, για την 1η Φεβρουαρίου είναι η ετήσια σύνοψη του προηγούμενου έτους, δηλαδή 1η Φεβρουαρίου είναι του έτους νη πλην 1 που θα πρέπει να παρουσιαστεί από τις αρχές. Και θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τις δικές μας ε, προτάσεις, ζητούμε να υπάρξει μια αιτήσια δήλωση ε, αξιοπιστίας όσον αφορά τα μία κοινή ε, επιμερισμένη διαχείριση. Και αυτή η κοινή, η δήλωση θα υπογράφεται από την αρμόδια αρχή που είναι διαπισταυμένη στι χώρε μέλη. Δεν θα υπογράφεται σε πολιτικό επίπεδο βεβαίω και ακού, άκουσα πολύ καλά τα όσα είπε ο κύριος Χάουζερ και θα έλεγα ότι πράγματι είναι μια, είναι μια πολιτική συζήτηση βάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει στο επίπεδο της αρχής διαχείρισης αυτή η δήλωση αξιοπιστίας θα υπογράφεται Ίσως στη συνέχεια θα ε, ε, ε, θα αποφασιστεί ποιο θα υπογράφει σε πολιτικό επίπεδο, αυτό δεν θα συμπεριλαμβάνεται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Και ο καθηγητή Δημαρτίνο να απαντήσει σε άλλε και άλλε ερώτησει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόβλημα είναι το εξή. Ανάγκη ερμηνεία του 317. όπω είπα και πριν, με προσφυγή σε ένα κριτήριο μη καταγράμμα ερμηνεία, λογική ερμηνεία. Ξεκινάμε την υπόθεση. Ευθύνη της Κομισιόν στην εκτέλεση του προπολογισμού. Βέβαια, με μια σχέση συνεργασίας που το άρθρο δεν το αναφέρει ρητά. Η σχέση με τα άρθρα 310, 325 και 122 με μορφές παρέμβασης εκ μέρους της Κομισιόν στη συνεργασία με τα κρατη με γενικό σεβασμό των κανόνων χρηστής οικονομικής διαχείρισης απαιτεί τον εντοπισμό του κατά πόσον το κράτος τηρεί αυτό που πρέπει να τηρεί χρειάζεται παρέμβαση. Και το πρόβλημα είναι το εξή. Σε ένα κράτο δικαίου η παράβαση μιας υποχρέωσης, η μη συμμόρφωση, σημαίνει κυρώσει για την μη τήρηση αυτή. Η συνθήκη όμως αφήνει κάπως το θέμα ανοιχτό σχετικά με το την ανάγκη η Ένωση στην περίπτωση μη συνεργασίας με το κράτος μέλος και από την άλλη μεριά την ανάγκη σεβασμού της εθνικής επικυριαρχίας εκ μέρους των οργάνων της Ένωσης. Αν όμως, ως υπόθεση, όπως είπε πριν σε μια παρέμβαση συνάδελφος η μη τήρηση προέρχεται από συμπεριφορά του κράτους θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει νομοθεσία που να δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να κάνει και έλεγχο να έχει τη δυνατότητα παρέμβασης που αντικειμενικά να αφαιρεί από το κράτος τη δυνατότητα να διαπράττει μια τέτοια πράξη μη τήρησης, μια πράξη που γίνεται μέσα στα, στον γεωγραφικό του χώρο. Ο Σνέφος Ριβελίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάτι δεν καταλαβαίνω εδώ για το περιθώριο σφάλματος ή ορίζεται και το δεχόμαστε γιατί θεωρούμε δεδομένο ένα περιθώριο σφάλματος ή η μελέτη θα πρέπει να έχει σαν στόχο το γιατί υπάρχει σφάλμα. Εδώ κάτι δεν πάει καλά με τη συζήτηση αυτή. Και σε σχέση με αυτά που μας είπε η Κομισιόν, δηλαδή ή δεχόμαστε ένα συγκεκριμένο ποσοστό ασφάλματος και προχωρούμε ή θα πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία του ασφάλματος και όχι το ποσοστό ασφάλματος. Ο κύριος Χάουζερ. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω σε κάποια σε κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν, όσον αφορά αυτό που είπε η Κομισιόν για τον ήμιον 1 ή ήμιον 2. Πράγματι, τα έγγραφα που υποβάλλονται στις 15 Φεβρουαρίου είναι νήμιον 1. Αναφέρονται στο έτος νήμιον 1. Οι έλεγχοι όμως στα έγγραφα αυτά αναφέρονται στο οικονομικό έτος νήμιον 2. Και εδώ υπάρχει το κενό ανάμεσα σε αυτό που λαμβάνουμε από το ελεγκτικό συνέδριο στην δήλωση εξοπιστία και αυτό που παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση. Όσον αφορά το περιθώριο ανοχής, όσον αφορά ε, τα σφάλματα. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Ριβελίνη, είναι μια πολιτική απόφαση, το δέχομαι. σε ποιες περιπτώσεις το κοινό θα ε, διαμαρτυρηθεί. Ε, και σε ποιες περιπτώσεις θα, τα, θα αφήσει τα ε, λάθη να περάσουν. Αλλά αυτό δεν φτάνει στη, στη ρίζα του προβλήματος. Πού δημιουργείται το λάθος. Ε, εάν δεν γνωρίζουμε τους λόγους δεν μπορούμε να να αποφασίσουμε αν ένα λάθος ε, είναι ανεκτό ή όχι. Ε, εντάξει, μιλάμε για ναι, εντάξει, ένα εκατομμύριο, δέκα εκατομμύρια λάθος, τρία εκατομμύρια λάθος. Όταν φτάνουμε στο δισεκατομμύριο αρχίζει και γίνεται προβληματική η κατάσταση. Όσον αφορά το ερώτημα... Τι κάνει ο εξωτερικός οικονομικός έλεγχος. Ενεργεί ε, ενάντια στα συμφέροντα του ε, ίδιου κρατούς μέλους. Με άλλα λόγια, ο ε, εξωτερικός λογιστικός έλεγχος είναι διατεθειμένος να εξετάσει τα λάθη που πραγματοποιούνται στην ίδια του τη χώρα. Εάν έχουμε ένα αυτόματο σύστημα κυρώσεων, τότε μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν ρωτήσουμε τον απαταιώνα τι ε, ποινή θα ήθελε, πόσο μάλλον αν δεν θέλει καμία, τότε δεν μπορείτε να ε, περιμένετε σωστή απάντηση. Το ίδιο ισχύει και με τα κρατη και για όλους μας ισχύει. Αν δεν το πετύχετε αυτό, ξεχάστε τα όλα. Όσον αφορά τα ελεγκτικά συνέδρια, ε, ή το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, ναι, κάποια κάποια ζώα, είναι ανώτερα από κάποια άλλα, ε, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικές, ε, υποχρεωτικούς κανόνες. Ποιος ελέγχει και ποιες ερωτήσεις θα πρέπει να απαντώνται. Δεν μπορεί να πει κανείς έτσι ότι διασφαλίζεται σε ένα κράτος μέλος εφόσον είναι θετική η δήλωση αξιοπιστίας ότι δεν γίνονται λάθη στο κράτος μέλος αυτό και έτσι φτάνουμε πάλι στο σύστημα κυρώσεων. Η Κομισιόν όταν κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους που πρέπει να τους κάνει, θα πρέπει να τους κάνει, εάν δείξουν λοιπόν ότι οι δηλώσεις αξιοπιστίας ή ε, οι εκθέσεις του εξωτερικού ελέγχου έχουν λάθη, ε, θα πρέπει να υπάρχει αυτόματο σύστημα κυρώσεων και θα πρέπει να πονάει τόσο πολύ η κύρωση ώστε ένα κράτος μέλος να σκεφτεί ε, δύο φορές αν θέλει να επιτρέψει ένα τέτοιο λάθος στη χώρα του. Αλλά Υπάρχει μια παρηγοριά τουλάχιστον για τα κράτη-μέλη. Τη στιγμή που ένα κράτο-μέλο ανακαλύπτει μόνο του ένα λάθο και εντό λογικού χρονικού διαστήματο διορθώνει το λάθο, δεν θα χάνει ε, πόρους που θα μπορεί να τους διατηρήσουν και πιστεύω ότι ήδη σήμερα λοιπόν είναι δυνατόν να αρχίσουμε να ψάχνουμε, ε, να βρούμε τα λάθη ε, χωρίς να ε, πονέσει το ίδιο κράτος μέλος. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόστοκ από το Ελεκτικό Συνέδριο προτού να φτάσουμε στη γενική συζήτηση. Όπως ε, είπε ο Γενικός Διευθυντής, ε, οι πολιετής ε, διορθωτικές εκθέσεις της Κομισιόν δείχνουν ότι υπάρχει ε, κάποιο κενό. Και ναι, η Κομισιόν λέει εντάξει μη σα νοιάζει το περιθώριο λάθους, ε, στο μέλλον θα το διορθώσουμε. Τρεις παρατηρήσεις από το ελεγκτικό συνέδριο. Σε αρκετές αιτήσεις εκθέσεις έχουμε πει ότι Περιμένουμε αξιόπιστα ε, στοιχεία για τα θέματα αυτά. Περιμένουμε ακόμα όμως. Δεύτερον, η περσινή ετήσια έκθεση εντόπισε κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα διόρθωσης των διαφορετικών ταμείων όπου κάποια μη επιλέξιμα προγράμματα ε, αντικαταστάθηκαν από κάποια εξίσου μη επιλέξιμα προγράμματα. Δεν ήταν πολύ καλή η διόρθωση αυτή. Και τρίτον, νομίζω ότι είναι αλήθεια ότι η βασική μορφή δράσης της Κομισιόν δεν έχει να κάνει με επιστροφή ε, χρημάτων που δόθηκαν ε, λανθασμένα, αλλά στην ανάκτηση χρημάτων από τους φορολογούμενους των κρατών μελών. Το να, ε, ανακτά όμως πόρους από τους ε, φορολογούμενους ε, δεν είναι μηχανισμός διόρθωσης ε, λαθών, είναι μηχανισμός κοινωνικοποίησης των λαθών, δηλαδή να μοιραζόμαστε πιο πολλοί άνθρωποι τα λάθη της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν δεν έχουμε άλλες παρεμβάσεις, ας περάσουμε στην επόμενη τμήμα της ακρέασης. Ο κύριος Μπόστοκ Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εμπειρίες από τα τρέχοντα δημοσιονομικό κανονισμό και την ανάγκη αναθεώρησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ τις Επιτροπές Προπολογισμού και Ελέγχου του Προπολογισμού για την πρόσκληση στην ακρόαση αυτή. Με ενδιαφέρον άκουσα τους σημερινούς ομιλητές για το τι ευχαρίστηση και τι απογοητεύσεις έχουν όταν δουλεύουν με τους τρέχοντα δημοσιονομικό κανονισμό και αυτό μας θυμίζει ότι το να ορίσουμε κανόνας στοιχίζει και το κόστος βαρύνει κυρίω όχι αυτός οι οποίοι προτείνουν τους κανόνες και επειδή το ελεκτικό συνέδριο τα ξέρει όλα αυτά γι' αυτό είδαμε και εμείς το κόστος που φέρουν οι δικαιούχοι σε εκθέσεις όπως αυτό για το έξυπνη ενέργεια την Ευρώπη πριν από μερικά χρόνια και επειδή ακριβώ το έχουμε επίγνωση στο γεγονότος, γι' αυτό ζητήσαμε απλούστευση των κανόνων. Και πιο πρόσφατα στη γνωμοδότησή μα 1 του 2010 για του κινδύνους και τις προκλήσεις για την Ένωση. Ε, ήμουν κάπω αγενής λοιπόν με την Κομισιόν, τώρα θα πω και κάτι υπέρ της Κομισιόν. Τους ευχαριστώ στην Κομισιόν γιατί τη βάλανε στο έγγραφο της δημόσιας διαβούλευση μερικά ωραία, ωραίες ερωτήσεις και ωραίες προτάσεις όπως επιλογές για πλούστευση να αυξημένη η χρήση των πληρωμών κατά αποκοπήν και οι επιδοτήσεις να εξαρτώνται από την επίδοση. Ωστόσο πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το να αλλάξουμε τον δημοσιονομικό κορονισμό είναι μόνο ένα τμήμα μιας διαδικασίας μείωση του βάρους για τους δικαιούχους και μέρος της διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας της ε, δαπάνης της Ένωσης. Πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορές, αποτελέσματα, νομικά εργαλεία. Πρέπει να μετρήσουμε την πρόοδο της απλούστευσης και όπως είπε πιο πριν ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι, οι βασικοί κανόνες που καλύπτουν τις δαπάνες της Ένωσης συχνά εμπρέχονται στις γενικές σελίδες του δημοσιονομικού κανονισμού αλλά στις λεπτομέρειες του κανονισμού κατά τομέα και φαίνεται να υπάρχουν ορισμένα εθνικά προβλήματα όπως ακούσαμε. Χώρες που κάπως τις ξέρω. Ίσως μερικά από τα εθνικά αυτά προβλήματα θα πρέπει κυρίως να ε, αντιμετωπιστούν στη συγκεκριμένη χώρα κάθε φορά. Βέβαια αυτό δεν είναι λόγος να είμαστε απεσιόδοξοι για την προοπτική απλούστευσης. Ο μεγάλος τομέας όπου ήδη η απλούστευση έγινε είναι η γεωργία. Το σύστημα των, ε, το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης πληρωμών είναι πιο απλό. Είναι πιο απλό από το προηγούμενο και το ποσοστό σφάλματος που διαπιστώνει η Κομισιόν είναι όλο και πιο μικρό. Αλλά σε άλλους τομείς δαπάνης επιπλέον απαιτήσει σε βάρος των δικαιούχων πολλές φορές είναι εναλλακτική λύση ως προς την απλούστευση των κανόνων ή προς απλούστευση του ίδιου του, του, της, της μεθόδου. Και η, η εμπειρία που έχουμε από το ελεγκτικό συνέδριο και που ακούσαμε σήμερα δείχνουν ότι αυτά είναι σε βάρος των δικαιούχων. Κύριε και κυρία Πρόεδρε, ας επανέλθω στο σημερινό μας θέμα που είναι η μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού. Προτείναμε η διαχείριση των προγραμμάτων δαπάνη στο μέλλον να έχει σαν στόχο την επίτευξη στόχων και όχι έλεγχο του input των εισρώων. Επίσης είπαμε η Κομισιόν να αξιολογεί όλα τα στοιχεία κόστους στα προγράμματα αυτά ακόμα και αυτά που επιβάλλονται στα κράτη-μέλη και στους δικαιούχους και το συνέδριο με ευχαρίστηση βλέπει ότι πολλές από τις προτάσεις μας αντικατοπτρίζονται στις προτάσεις της Κομισιόν που μόλις τώρα πήραμε και τις μελετάμε με ενθουσιασμό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, την τελευταία δεκαετία οι τροπολογίες για το δημοσιονομικό κανονισμό έγιναν στα πλαίσια, στα πλαίσια. Τώρα ξεκινάμε με πιο μεγάλες φιλοδοξίες και όπως πολλοί ευρωβουλευτές μας το θύμισαν γίνεται μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο ευθυνών. Εμείς περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα ως παρατηρητές, παραδείγματος χάρη, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι πρόοδος θα γίνει στο ανεκτό κίνδυνο ή ανεκτό σφάλμα. Θα είναι μηδενική ανοχή. Εσείς κύριε Πρόεδρε πριν από δύο μισή ώρες αναφερθήκατε σε αυτό, είπατε μηδενική ανοχή. Επίσης περιμένουμε και την συζήτηση που θα γίνει και ως συμμετέχοντες, διότι θα δώσουμε γνωμοδότηση στην πρόταση, θα παίξουμε το ρόλο μας πλήρως προκειμένου να, υπάρχουν, να υπάρξουν πιο απλοί κανόνες με μεγαλύτερη εστίαση στην απόδοση και επίδοση προς όφελος των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπόστοκ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τώρα το λόγο στους δύο εισηγητές της Επιτροπής Προπολογισμών και Ελέγχου Προπολογισμού, κύριε Γκρέσλε και Ριβελίνια. Η κυρία Γκρέσλε είναι μέλος και στις δύο επιτροπές. Επειδή ο δικαστής, η δικαστής Πιτσιρίλο δεν μπόρεσε να έρθει, θα μας μιλούσε για τη διαχείριση και εθνικές δηλώσεις των κρατών μελών και υποχρεωτικά περιεχόμενα πιθανών νομικών διατάξεων Επειδή έχουμε χρόνο, οι εισηγητές θα μπορούσαν να αναφερθούν στο σημείο αυτό, αν θέλουν. Αρχίζουμε με την συνάδελφο Γκρέσλε. Ε, συγγνώμη, εδώ υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα με το μικρόφωνο μου. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω κάποιες, ε, κάποια μικρά σχόλια. Αλλά τελικά μου είπατε ότι θα πρέπει να αντικαταστήσω ε, τον εισηγητή που δεν ήρθε. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση η οποία παρουσιάστηκε εδώ. Είναι πραγματικά εξαιρετική. Και πραγματικά ε, καλώς ήρθατε στο κλαμπ. Γιατί πραγματικά θα έδινα πολλά αν αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει το 2006 γιατί τότε ήταν σε με πολλούς κόπους να κάνουμε κάποιες διευκολύνσεις. Για να σας δώσω ένα σύντομο ιστορικό. Και η κυρία Τότ μίλησε σχετικά για τις, σημαντικά, για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Η τελευταία μεταρρύθμιση το 2006 ήταν μια μεταρρύθμιση που έκανε η Επιτροπή για τον εαυτό της και οι διευκολύνσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή χρησιμεύουν κυρίως στην ε, Κομισιόν και το θέμα των δικαιούχων τότε δεν είχε τεθεί. Βεβαίως έγιναν κάποιες ε, βελτιώσεις ούτως ώστε η Επιτροπή να διαμορφωθεί σαν μια υπηρεσία φιλική προς τον πελάτη. Λοιπόν, μας παρουσιάστηκαν τώρα κάποια κομμάτια των νέων μεταρρυθμίσεων όπου συλλαμβάνονται κάποια στοιχεία των παλαιών ιδεών αλλά υπάρχουν και εντελώ καινούργιες ιδέες. Χαίρομαι λοιπόν που επιτέλους έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για μια νέα διαμόρφωση του δημοσιονομικού κανονισμού. Αλλά αυτή η νέα διατύπωση δεν θα χρησιμοποιήσει σε τίποτα εάν άλλα τμήματα της Κομισιόν τελικά επιβάλλουν κάποιους, νέους, κάποιους άλλους κανόνες για τα ειδικά ταμεία που αντιβαίνουν ε, στον κανονισμό αυτό και αυτό είναι ακριβώς που φοβάμαι και αυτό που πραγματικά με απογοητεύει συνεχώς να διαπιστώνουμε ότι είμαστε ανίκανοι να αντιλήσουμε διδάγματα από τις εμπειρίες μας. Γι' αυτό είναι κατεπίγουσα παράκληση και προς τον Επίτροπο να μην γίνει κάτι τέτοιο γιατί αν δεν το πετύχουμε νομίζω ότι θα πάει χαμένη όλη αυτή η καλή συνεργασία μεταξύ μας. Τώρα, ε, η Κομισιόν στις προτάσεις της πολλές προτάσεις των Επιτροπών του Κοινοβουλίου. Τώρα, το, θέμα, το ερώτημα ποιο είναι τμήμα της ερώτησης και ποιο είναι τμήμα της απάντησης, το απαντώ ως εξή. Εμείς έχουμε ε, ζητήσει πολλές ε, διευκολύνσεις ε, και βελτιώσεις από το τμήμα, από το τομέα της, από το τμήμα της έρευνας και πρόκειται να εξετάσουμε αυτά τα πολύ λεπτομερή κείμενα. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν και οι κανόνες εφαρμογής και νομίζω ότι αυτό διευκολύνει από τη μία την εργασία μας, από την άλλη τη γιατί είναι υπερβολικό όγκο τη εργασία. Έχουμε 480 σελίδε, εφαρμοστικέ διατάξει. Αυτό το είπε και η κυρία Πρόεδρο. Έχουμε τρει διαδικασίε και. Ε, ε, η πρώτη αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα γίνει τελευταία δηλαδή θα ασχοληθούμε ε, καταρχήν με, τα, με άλλα πράγματα. Η πρώτη διαδικασία αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Το δεύτερο ε, είναι το recast και το τρίτο είναι η τροποποίηση του κανονισμού σε σχέση με τη συνθήκη Λισαβόνας. Δηλαδή αυτό που τελικά θα εφαρμόσουμε, το οποίο μπορεί να περιμένει περισσότερο από τα άλλα. ο κ. Ριβελίνη και εγώ προσπαθούμε να δούμε ποια άρθρα κατ' ουσία θα πρέπει να γίνουν αντικείμενα επεξεργασία στο πλαίσιο αυτών των τριών διαδικασιών. Και θα πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι ιδιαίτερο εύκολο, γιατί αυτή την εργασία δυστυχώς δεν την έκανε η Επιτροπή. Σε τρεις διαδικασίες τελικά γίνονται αντικείμενα σε τρία διαφορετικά άρθρα. Το άρθρο 1, 49 και 23 με τα άρθρα αυτά συγγνώμη, ασχολούνται και οι τρει διαδικασίε, αλλά χωρί ε, η κάθε διαδικασία τελικά να μπορεί να επανέρχεται στην εργασία που έχει ήδη γίνει στο πλαίσιο τη πρώτερη διαδικασία. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αν δεν είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, τελικά τα αποτελέσματα θα είναι χάο, θα ξεσπάσει το χάος στο τέλος. Έχουμε το ζήτημα του υπολογισμού των, του κόστους για το προσωπικό, το ζήτημα των επιτοκίων κλπ. Επίσης μια εξέταση των μεθόδων βέλτιστων πρακτικών στις χώρες μέλη κλπ. Νομίζω αυτό το σημείο είναι καλό για μας. Παρόλο που εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση εν σχέση με το τι είναι βέλτιστες πρακτικές και το τι είναι απλούστατα άγνοια θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και να κάνουμε σχετικά πολλέ συζητήσει. Για παράδειγμα, τόσο είπε ο κ. Μίτσελ για τη Μεγάλη Βρετανία, μου κατέστησε σαφέ πόσο σύνθετο είναι αυτό, το πολύπλοκο αυτό το εγχείρημα, να θέλουμε με ένα ενίο σώμα κανόνων να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και καταλήγουμε στο ερώτημα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Επιτροπή Προπολογισμού και Ελέγχου του Προπολογισμού. Τι γίνεται με τι εθνικέ δηλώσει αξιοπιστία και άλλα θέματα ιδιαίτερα σημαντικά για μας. Η διαφάνεια, πραγματικά το ορόσημο της τελευταίας ε, ε, μεταρρύθμισης. Θεωρώ ότι η διαφάνεια είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Επιτροπής Μπαρόζο. Νομίζω ότι αυτή η Κομισιόν δεν με το θέμα αυτό, νομίζω ότι πραγματικά είναι ντροπή. Δεν γίνεται μνήα στο θέμα αυτό και αν δούμε την πληθώρα των δημοσιεύσεων στις χώρες μέλη που θα έπρεπε να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα εν σχέση με το ποιος παίρνει τα ευρωπαϊκά κονδύλια νομίζω ότι οι δημοσιεύσει αυτές θα πρέπει να βελτιωθούν και να γίνουν πιο ενιαίες και θα πρέπει εμείς ως Κοινοβούλιο να υποβάλουμε σχετικές προτάσεις. Τώρα, όσον αφορά το ανεκτό περιθώριο σφάλματος, θα ήθελα να πω ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν σήμερα είναι απολύτως δικαιολογημένα. Δεν νομίζω ότι Ε, δεν ξέρω, μπορούμε να σπαταλήσουμε για παράδειγμα ένα δισεκατομμύριο ευρώ ως ε, περιθώριο αποδεκτού σφάλματος. εδώ είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε, δηλαδή τι ακριβώς θέλουμε και πώς βλέπουμε τα πράγματα. Χωρίς τη στήριξη της Επιτροπής και των δύο Επιτρόπων αυτό δεν θα γίνει. Και θα ήθελα πραγματικά να ξέρω την ε, προεργασία της Επιτρόπου Προϋπολογισμού που φρόντισε ούτως ώστε οι εφαρμοστικές διατάξεις να συμπεριληφθούν ε, στην συναπόφαση. Έχουμε μια όπου υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία, για παράδειγμα τη διαδικασία του προπολογισμού ή ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός ε, είναι για πρώτη φορά στην απόφαση. Θυμάμαι την τελευταία μεταρρύθμιση όπου χρειαστήκαμε μισό χρόνο για να δούμε ποιον θα πρέπει να πάρουμε το μέρο μας για να πετύχουμε κάποια πράγματα. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή κλείπουν και μπορούμε να συγκεντρωθούμε στα περιεχόμενα. Κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα πράξουμε και νομίζω ότι αυτή είναι μια ευκαιρία που έχουμε και που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ούτω ώστε να μεριμνήσουμε για να διευκολυνθούν οι ροές των χρημάτων αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρηθεί η ποικιλομορφία, κάτι που είπε ο κ. Ματζίστρης. Δηλαδή, ε, τι γίνεται με την ε, επινοητικότητα των εγκληματιών που, των κακοποιών που παίρνουν χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα πρέπει να το δούμε αυτό και θα πρέπει να συντονίσουμε τις ενέργειές μας ούτε ώστε το 2011 να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και η πρώτη ανάγνωση μέχρι το τέλος του χρόνου να προγραμματιστεί και μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου έτους να προχωρήσουμε να προγραμματεύσουμε το Συμβούλιο ούτε ώστε ήδη το 2012 να ξέρουμε τι έχουμε να περιμένουμε από το δημοσιονομικό κανονισμό. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη γραμματεία του σώματος γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν δυνατό να γίνει αυτό το ε, έργο και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Μαγιόφσκα και ελπίζω να συνεργαστεί ε, μαζί μας και στο μέλλον. Ε, είπα στο δικό μου βοηθό να μην κάνει επικίνδυνα σπορ, να κάθεται στον καναπέ του και να φροντίζει τον εαυτό του γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το έργο και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να μας ε, δώσουν τις ιδέες τους, γιατί είναι μια πραγματική ευκαιρία να δούμε το έργο αυτό σαν μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παραμείνετε σε επαφή μαζί μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να πω θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ιδιαίτερως ε, θέματα παραμένουν εκρεμή, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Τόσα έχουμε στα χέρια μας δεν είναι ικανοποιητικά, γιατί αφορούν ή μάλλον ε, ε αναβάλλονται οι δηλώσεις αξιοπιστίας για το 2015 το 14 να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και το 15 να είναι έτοιμες. Και νομίζω δεν θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό, τέτοια αναβολή. Και δύο επιτροπές καλούνται να συμπεριλάμβουν τα θέματα που θεωρούν σημαντικά. Εμείς θα το πράξουμε. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους το θέμα αυτό που μας απασχολεί που θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό ε, να το προσεγγίσουν με την απαιτούμενη υπομονή. γιατί το χρειάζονται οι συγητές. Δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται οι συγητές να αφυπνίσουν κάθε φορά τον ενθουσιασμό των ακροατών τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκρέσλε και ο άλλος συζητητής μας, ελέγχο προπολογισμού, ο κύριος Ρεβελίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τους συμμετέχοντες για όλες τις εκθέσεις που ακούσαμε. Πολύ ενδιαφέρουσες και δείχνουν για μια φορά ακόμα που η πανεπιστημιακή και η ειδική του τομέα μπορούν να βοηθήσουν τους νομοθέτες το θέμα μας αυτό είναι πολύ φιλόδοξο. Μία αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού με προοπτική της Ευρώπης 2020 απασχολεί δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πολλά θέματα συζητήθηκαν σήμερα και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον οι παρεμβάσεις που αφορούν τη δική μας Επιτροπή για την οποία είμαι και εισηγητής. Ιδιαίτερα εκτιμήσα την έκθεση του Δ. Ντόρτι που αναφέρθηκε στα υπέρ και τα κατά της τελευταίας αναθεώρησης του 2005 και τόνισε την επιτάχυση των διαδικασιών πληρωμών ε, κονδυλίων της Ένωσης με καλύτερη πληροφόρηση. Επίσης, το πώς μειώθηκε το διοικητικό άχθος όσον αφορά τις, ε, τους διαγωνισμούς και τις προσφορές. Βέβαια, παραμένουν πολλές γκρίζε ζώνες, όπως η πρόσβαση στα κονδύλια, που συχνά αποκλείει πολλούς λόγω του ότι απαιτούνται πάρα πολλά ε, κείμενα και υπάρχει και διαφάνεια. Μια νέα νομοθεσία δημοσιονομικού χαρακτήρα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλούστευση των διαδικασιών έτσι ώστε ο πολίτες, οι διάφοροι οργανισμοί να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τη σωστή χρήση, λογιστική χρήση του κάθε ευρώ που δαπανάτε και ταυτόχρονα επιτρέπουμε εκατομμύρια πολίτες να μην γνωρίζουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η Ευρώπη. Και λόγω του υπερβολικής γραφειοκρατίας να παρεμποδίζονται στο έργο τους. Αυτό οδηγεί σε δημοκρατικό έλλειμμα που εμποδίζει μια αρμονική ανάπτυξη και έναν πιο δίκαιο επιμερισμό στη χρήση των κοινωτικών κονδυλίων. Όπως επίσης μπλοκάρει ιδέες και πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν. Βέβαια, η παραβολική γραφειοκρατία οδηγεί και σε απάτες. Επίσης εκτίμησε αυτά που είπε, ιδιαίτερα αυτά που είπε ο καθηγητής Δεμαρτίνο, ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα δύσκολο θέμα υποχρεώσει των κρατών μελών στην εφαρμογή του, του προπολογισμού και τόνισε ότι το άρθρο 317 ως έχει είναι και υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών αλλά πέραν του ελέγχου έχει λόγο ύπαρξης σε κοινή αντίληψη της κοινωνικής ευημερίας που εξασφαλίζεται μέσω και χρηματοδότησης με κοινοτικά κονδύλια. Άλλο θέμα, περίπλοκο και αυτό, πολύ ενδιαφέρον όμως, που θα το κάλυπτε η κυρία Πιτσιρίλου που δυστυχώς δεν ήρθε, είναι η κοινή διαχείριση των εθνικών δηλώσεων από τα κράτη-μέλη. Η εισαγωγή υποχρέωσης εθνικών δηλώσεων διαχείρισης που θα πρέπει να καταθέτουν όλες οι χώρες είναι η υπέρβαση της ετήσιας σύνθεσης που δυστυχώς απέδειξε ότι έχει περιορισμένη προστιθέμενη αξία γιατί η νομική βάση ήταν ανεπαρκής. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν, η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού πιο συγκεκριμένα, ανέκαθεν υποστηρίζουμε τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης και μια μελέτη της αιτήσιας σύνθεσης να γίνεται μια μελέτη που έγινε το 2009 απέδειξε ότι αυτό είναι απόλυτη ανάγκη να γίνει με βάση αυτή τη μελέτη η υποκατάσταση της αιτήσιας σύνθεσης με εθνικέ δηλώσεις διαχείρισης θα έχει ιδιαίτερα θετική επίπτωση στην ποιότητα των πληροφοριών που θα είναι πιο πλήρες και πιο αξιόπιστες. Τέλος, Ευχαριστώ τον ε, Αντιπρόεδρο του Γερμανικού Ελεκτρικού Συνεδρίου, τον Δ. Χάουζερ, ο οποίος με μια πολύ σαφή παρουσίαση που μας έκανε αναφέρθηκε στο θέμα της αξιοπιστίας στα ομοσπονδιακά συστήματα, ιδιαίτερα με βάση το άρθρο 53β του Δημοσιονομικού Κανονισμού της Ένωσης. Συγκεκριμένα, προσωπικά βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση να υπάρχει ένα DAS, μια δήλωση αξιοπιστίας κατά κράτος διαφοροποιημένη και κατά τομέα επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματική όσον αφορά την γεωργική πολιτική. Τέλος, ευχαριστώ και τη Σάφο Γκρέσλε με την οποία έχουμε δώσει από κοινού πολλές μάχες στην Επιτροπή μας και τους δύο πρόεδρους και τους βουλευτές που μίλησαν και τους εμπειρογνώμονες και πάλι. Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στον καθηγητή Μπόστοκ ο οποίος με σύντομη παρέμβαση τόνισε ακριβώς την ανάγκη της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού για να έχουμε δημοσιονομικούς κανόνες πιο απλούς και πιο εστιασμένους στο αποτέλεσμα και μερικά πολιτικά σχόλια. Γιατί, Γιατί είμαι πολιτικός. Είμαστε πολιτικό όργανο εδώ. Δημοκρατικά εκλεγμένο. Έχουμε την υποχρέωση πολιτικών αξιολογήσεων. Τι σημαίνει αυτό. Ναι, να απλουστεύσουμε τους γραφειοκρατικούς κανόνες για να αποφύγουμε απάτες. Ναι, ένας πιο καλός έλεγχος για να αποφύγουν διάφορες συγχύσεις κλπ. Αλλά για μας αυτό είναι ένα δευτερεύον τμήμα της δουλειάς μας. Γιατί αυτή τη δουλειά είναι να την κάνουν τα ελεγκτικά όργανα. Οι δικαστές, οι λογιστές, εμείς πιο σημαντική είναι η δουλειά μας και πιο δύσκολη να καταλάβουμε για όλα τα κοινωτικά κονδύλια να χρησιμοποιούνται γρήγορα και σωστά και στο σωστό χρόνο. Γιατί σε μια εποχή κρίσης των αγορών και παγκοσμιοποίησης ο χρόνος μετράει απόλυτα αν ένα κονδύλι δοθεί καθυστερημένα δεν μετράει. Όλοι, όλοι είπα πριν, κρίμα που σε μια περίοδο κρίσης να υπάρχουν κονδύλια που να μην χρησιμοποιούνται. Να καταλάβουμε πώς θα χρησιμοποιούνται στα σωστά κεφάλαια τα κονδύλια, αυτό είναι ε, έργο δικό μας, σημαντικό έργο. Να χρησιμοποιούνται καλά. Τι σημαίνει καλά, να χρησιμοποιούνται καλά τα, τα κονδύλια. Αυτό είναι το κέντρο της δουλειάς μας, μια ανάλυση του πώς και πού πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Σε κεφάλαια και σε τομείς όπου η δαπάνη θα είναι ικανοποιητική και χωρίς καθυστερήσεις. Διαφορετικά θα πλήξουμε την απασχόληση, την τεχνολογική καινοτομία, την ανάπτυξη της Ευρώπης. Και είναι αδίκημα αυτό παρόμοιο με τις απάτες. Και αν δεν πετύχω μία ισορροπία, οι απάτες και αν έχουμε και τις δαπάνες που δαπανώνται κακώς, θα έχουμε την κακή έκπληξη να διαπιστώσουμε ότι πιο μικρή μία ζημιά από τις απάτες από ότι η κακή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μετά τη Λισαβόνα λοιπόν και με περισσότερες εξουσίες που έχουμε Ας φροντίσουμε να δώσουμε μια σωστή απάντηση και να μην σταματάμε και μένουμε αποκλειστικά σε μάχες που είναι δίκαιες μεν, αλλά μικρότερες σημασίας και αξίας. Και επιτρέψτε μου να κάνω και μία μεταφορά. Εύχομαι Στο μέλλον το χρηματοκιβώτιο που είδαμε κάπου εδώ σε έμβλημα είναι από γυαλί. Να μπορεί κανείς να το δει και να το καταλάβει και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν τις περισσότερες ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Βελίνη. Η κυρία Τότ σύντομα έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο και νομίζω ότι είναι σημαντικό για, την, για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θα ήθελα να πω ότι καλό τα μέλη της Επιτροπής Προπολογισμού και Ελέγχου του Προπολογισμού να συμμετάσχουν επίσης στη διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου που βρίσκεται υπό εξέλιξη και όπου η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο. Είναι ο τριμερής διάλογος, ε, κομισιόν, χώρες μέλη, κοινεβούλιο και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών διάλογο στο πλαίσιο του οποίου συζητούμε το μέλλον συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτών των φορέων. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία να γίνει πράγματι μια διασύνδεση εφόσον η παρούσα αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα είναι η βάση του δημοσιονομικού κανονισμού για τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια διασύνδεση μεταξύ αυτής της διαδικασίας όπου προσπαθούμε να συνδέσουμε πολιτικές με τους ανεδειγμένους μηχανισμούς εφαρμογής. Να γίνει αυτή η σύνδεση μεταξύ αναθεώρησης και πολιτικής εφαρμογής. Και σύντομα στην, στην ε, κυρία Χαγ που είναι αντιπρόεδρος Επιτροπής Προπολογισμών. Ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι εγώ θα μιλούσα στο τέλος. Παρ' όλα αυτά θα είμαι σύντομη. Νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωινό. Δεν το είχα φανταστεί όταν ερχόμουν εδώ. Και θα πρέπει να σας το πω ειλικρινά. Πραγματικά ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα ρεθίσματα εδώ. Ακούσαμε τις νομικές αξιολογήσεις και είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε το πώ καμιά φορά μεταξύ δεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ορισμένοι τριγμοί. Γιατί φυσικά άκουσα ότι ο έπαινος του ελεγκτικού συνεδρίου ως προς την Επιτροπή ήταν ότι τουλάχιστον η Επιτροπή έθεσε τα σωστά ερωτήματα. Ένας κάπως ε, αμφισβητούμενος έπαινος. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνεργασία μεταξύ μας ούτως ώστε να έχουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή σωστούς κανόνες, καλή επικοινωνία επί των κανόνων αυτών, ενιαία ερμηνεία αυτών των κανόνων και αυτόματες Κυρώσει στην περίπτωση παραβίασης αυτών των κανόνων. Εάν μπορούμε να συνδυάσουμε όλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Σας εύχομαι μια καλή μεσημεριανή παύση. Τα μέλη της Επιτροπής θα τα δούμε γιατί στη συνέχεια θα έρθουν τα Εθνικά Κοινοβούλια και έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Καλό απόγευμα λοιπόν και καλή σας όρεξη ευχαριστώ Θα προσθέσω μόνο δύο τεινά. Στον πρώτο έτος εργασιών μας το βλέπουμε ήδη. Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία των θεσμικών οργάνων. για τη σωστή διαχείριση των ε, δημοσίων κονδυλίων με πρόβλεψη να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού συνεργάζεται και με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο και, και με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και το δεύτερο, όχι μόνο για τις κυρώσεις αλλά για την πρόληψη ενίσχυση των οργάνων εγγύησης με αυτονομία φυσικά θεωρώ σημαντική τη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου και η Όλαφ με τον διορισμό του νέου διευθυντή που θα γίνει σύντομα θα, δοθεί, θα δώσει μια νέα όθηση στην καταπολέμηση της απάτης και άλλη μια πρόκληση της συνθήκης της Λισαβόνας είναι η Eurojust και η σύσταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. με σημαντικό ρόλο. Συναντήσεις όπως σημαντική είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τέτοιες συναντήσεις, επαναλαμβάνω, αυξάνουν την επίγνωση των προβλημάτων και επειδή για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος που είναι πολύ εμπεριέχει μεγάλο κίνδυνο διαφθοράς, οικονομικής διαφθοράς. Το είπα εγώ, το τον άφερε και Γκρέσλε, επικίνδυνες μορφές οργανωμένου εγκλήματος επίσης. Μόνο αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταφέρουμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά, μόνο τότε θα καταδικάσουμε και θα εμποδίσουμε επικίνδυνες συμπεριφορές, αλλά και θα φροντίσουμε έτσι ώστε το δημόσιο χρήμα να χρησιμοποιείται για την οικονομική ανάπτυξη, για τη μείωση της ανεργίας και για να το πετύχουμε αυτό, πολλές φορές το ακούσαμε σήμερα, πρέπει τα ευρωπαϊκά όργανα να έχουν όλο και περισσότερο κύρος και φερεγγιότητα, άρα και δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης έναντι των κρατών μελών που δεν σέβονται την νομοθεσία σε βάρος όλων και των οργάνων της Ένωσης και των πολιτών. Σας ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ και τη συνάδελφο Χάουγκ και όλους τους άλλους συναδέλφους, εμπειρογνώμονες, στο Ελεκτικό Συνέδριο των Κομισιόν για την συμβολή σας στη σημερινή συνεδρίαση. Καλή σας μέρα. Εμείς θα ξανασυνεδριάσουμε στις 22 Ιουνίου.